Good afternoon, ladies and gentlemen. you this of the εργασιών μας, θα έχετε όλοι λάβει την διάταξη, Λέω Πρόεδρος. Ο κύριος Μίλτερ, έχετε τίποτε παρατηρήσεις επί της Όχι από βλέπω. Έχετε κάποια παρατήρηση όχι. Επομένω συγκρίνεται η μέση διάταξη. Έχω όμω και εγώ κάποιε προτάσει να σα υποβάλω. 18 ώρε. Ε, Συνήθω αυτό συζητείται με του συντονιστέ. Σε 6 ώρε, γιατί σε 6 ώρε. 6 ώρα συντονιστές, αλλά θα έχουμε αυτή τη συνάντηση για τον δημοσιονομικό κανονισμό. επομένω. στις 6 ώρα, στις 6, όσοι ενδιαφέρονται για τον δημοσιονομικό κανονισμό, μήπως είναι κλεισμένον, όχι, όχι. Οπότε θα συνδυάσει η μαδρία σας. Τώρα θα ήθελα τη γνώμη σας. σε σχέση με το τι θα, αν θα εγκρίνουμε ή όχι, την απαλλαγή του Συμβουλίου για το 2009. Κάποιο από το Συμβούλιο παρίσταται για να μας πει την άποψη του Συμβουλίου για άλλη μια φορά. Οπότε και στη συνέχεια εσείς μπορείτε να σχολιάσετε. Όχι. Επομένως, να αλλάξουμε τη μέση διαδέξη τόσο στις 11 η ώρα να ακούσουμε το Συμβούλιο και φυσικά να ζητήσουμε το Συμβούλιο να στείλει κάποιον. Ωραία. Συμφωνείτε. Αυτό είναι σε διάταξη. Τώρα, ανακοινώσει του Πρόεδρο. Πέραν των γλωσσών εργασίας της μήνυμα συνεδρίαση, βλέπετε στο κοκομπού info θα πρέπει να σας πω ότι δυστυχώς δεν θα έχουμε διερμηνία ε, προς τα ρουμανικά γιατί είναι άρρωστοι οι ρουμανοί διερμηνείς από ό,τι μας είπαν. Επομένως όποιος θέλει να ε, ακούσει την ρουμανική καμπίνα θα πρέπει να αναζητήσει τα ρουμανικά άλλο. Μεταδίδεται με το web streaming η συνεδρίασή μα. Προσέχετε τι λέτε. Οπότε τελειώσαμε σε αυτέ τι ανακοινώσει και πάμε στο σημείο 3 τη μεσή διατάξεω. Απαλλαγή 2010. Θα δώσουμε το λόγο στον εισηγητή για το θέμα αυτό που είναι ο κύριο Φιόλνερ. Έχετε το λόγο, συνέχεια. Σα ευχαριστώ πολύ. Λέει ο κύριο Φιόλνερ. Θα πρέπει να σα πω ότι κατά τη γνώμη μου ε, που ήταν πάρα πολύ διαφωτιστική η σχετική έκθεση παρά το ότι έχουμε όλα αυτά τα έγγραφα και πολλές φορές ε, κανείς αναρωτιέται αν ε, λένε πολλά ή δεν λένε τίποτα. Γιατί όταν έχουμε κάποια σύνοψη, τι γίνεται, η σύνοψη μήπως καμιά φορά αποκρύπτει, κάποια δεν τα αναφέρει. Αυτό είναι σημαντικό, θα πρέπει να αναφέρουμε. Οπότε και εγώ θα ήθελα σε σχέση με αυτό να σας πω ότι όλοι, εάν θέλετε, μπορείτε να διαβάσετε αυτό το κείμενο, να ενημερωθείτε. Όμως, θα ήθελα να ακούσω την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να μας πούν εκείνοι τι πιστεύουν. Οπότε και θα είναι ενδιαφέρον να διαπιστώσουμε Και Οπότε για να δούμε εμεί τι θα πούμε, θα πρέπει να ακούσουμε τι έχει να πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τέλεια, λέει ο Πρόεδρο, πάρα πολύ σωστή αυτή η πρότασή σα. Και τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχει το λόγο, κύριε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμοι κύριοι βουλευτέ, κυρίε και κύριοι. Να σας πω εγώ τι έγινε όσον αφορά το πεπραγμένα του 2010 για την ετησία έκθεση. Έχουμε την, τον ιστορικό έλεγχο από το 2010, αλλά δεν μπορέσαμε ε, έγκαιρα ε, να σας την στείλουμε για να την έχετε για τη σημερινή συνάντηση. Οπότε και εγώ να σας πω δύο λόγια. Όμως ε, είμαι έτοιμος για να το συζητήσουμε όταν τον ε, Δεκέμβριο έρθει για την απαλλαγή να το συζητήσουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η έκθεση και είναι εδώ πέρα ένα μέσον ε, ε, δημοκρατικού ελέγχου, λογοδοσίας, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό όσον αφορά τη διαχείριση των πόρων και την επιλέξη των στόχων. Επίσης όμως θα πρέπει να δούμε κατά πόσον θα μπορούσαμε να έχουμε ιστορικούς ελέγχους. Επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον μας σε αυτές τις ε, αιτήσει ε, εκθέσεις δραστηριότητα και σε σχέση με το τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε την κατάσταση. Κοινοβούλιο, Συμβούλιο και Ελληνικό Συνέδριο είναι συναρμόδιοι και ε, επίσης αυτές οι εκθέσεις είναι και στο Ευρώτα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, μπορεί να έχει πρόσβαση αν θέλει σε αυτό το site. Οπότε έχουμε 17 επιφυλάξεις στην έκθεση του 2010 ενώ το 2009 είχαμε 20 επιφυλάξεις. 15 από αυτές ε, μεταφέρθηκαν από τον προηγούμενο χρόνο και έχουμε δύο τελείως καινούργιες. Πρώτα-πρώτα έχουμε την επιφύλαξη από τον Γενικό Διευθυντή για την αλλαγή του κλίματος και κατόπιν έχουμε τις κυβερνοεπιθέσεις στο σύστημα ε, Δεκεμβρίου 2010 και Ιανουαρίου 2011. Η δεύτερη νέα επιφύλαξη είναι αυτή που υπέβαλε ο επικεφαλής της ε, εκτελεστικής υπηρεσίας όσον αφορά την διαχείριση του πολιτικού προγράμματος. Μετά από τα ελληνικά ε, συνθήκες συνέργειες είχαμε 25% των ε, ε, επιφυλάξεων των περσινών που θα μπορούσαν τώρα να αρθούν. Η άρση αυτών των επιφυλάξεων όμως δεν θα πρέπει να θεωρείται ως χαλάρωση της ποιότητας της διαχείρισης και του ελέγχου. Όποτε έχουμε άρση της επιφύλαξης, όλα αυτά γίνονται μόνο αν έχουμε κατάλληλες πληροφορίες, ούτως ώστε να διαπιστώνεται ότι το πρόβλημα αντιμετωπίζεται επί τόπου. Σε αυτή την περίπτωση εδώ έχουμε συγκεκριμένε πληροφορίε ότι τα λάθη έχουν μειωθεί και ότι τα συστήματα ελέγχου έχουν αναβαθμιστεί. Οπότε και οι υπηρεσίε μας όλα αυτά τα έχουν επαληθεύσει και σε πολιτικό επίπεδο. Αυτή η έκθεση, η συνθετική, ε, περιέχει επίσης τα εξής τρία στοιχεία. Πρώτα-πρώτα, την ευθύνη, ευθύνη των κρατών μελών για, το, για την αποτελεσματική διαχείριση των κοινοτικών πόρων και την κοινή διαχείριση. Ακριβώς επειδή έχουμε αυτές, αυτή τη συνυπευθυνότητα που προβλέψει τις Λισαβόνες εμείς λέμε ότι θα πρέπει να ενδυναμωθούν τα αισθήματα ελέγχου και ιδίως το πρώτο επίπεδο των ελέγχων διαχείρισης. Πριν οι αξιώσεις, οι απαιτήσει για τους ελέγχους πιστοποιηθούν. Το 2010 έχουμε διακοπές που διακόπησαν του ύψους των 2,4 δις ευρώ και για ανασταλήσεις πληρωμές ε, αυτό γίνεται όταν βλέπουμε ότι υπάρχει σημαντική ε, έλλειψη, σημαντική υστέρηση όσον αφορά τον έλεγχο και τη διαχείριση των πόρων. Εμεί θα συνεχίσουμε αυστηρά την εποπτική μα λειτουργία και απευθυνόμαστε στα κράτη-μέλη και του ε, ζητάμε να αντιμετωπίσουν τι αδυναμίες του όσον αφορά τη διαχείριση και τον έλεγχο. Και αυτό, εάν έχουμε ε, όποτε πρέπει αυτές τις αναστολές, τις διορθώσεις, τις διακοπές των πληρωμών. Η πρότασή μας όσον αφορά τις αιτήσει δηλώσεις της διαχείρισης γίνονται επί τη βάση του δημιουργικού κανονισμού και για την ε, κοινή διαχείριση που είναι ο ακρογωνίος ε, λίθος ε, του, δημοκρατικού ελέγχου και της λογοδοσίας της υποχρεωτικής των κρατών μελών παρακαλώ να εγκρίνετε αυτή μας την, την πρόταση γιατί κατά δεύτερο λόγο αναγνωρίζουμε τη δυσκολία αυτών των ε, περιπλόκων κανόνων για τους ελτόμενους. Θα πρέπει επομένω να απλουστεύσουμε τους κανόνες, ούτω ώστε να έχουμε αναθεώρηση του δημοσιογού κανονισμού και τώρα θα πρέπει να ολοκληρώσουμε αυτές τις απλοποιήσεις ε, και στην ε, νομοθεσία ανά θέμα. Ήδη έχουμε διατυπώσει προτάσεις στα πλαίσια δημοσίου κανονισμού, ούτω ώστε να μπορέσουμε να μειώσουμε τα λάθη και έτσι να γίνει ε, το μοναδικό κόστος να συρρυκνωθεί, να δούμε τι θα γίνει ε, με τα κατακοποκοπή ποσά και επίσης έχουμε κάποιες φιλόδοξες προτάσεις για να απλουστευτεί η διαχείριση όσον αφορά την έρευνα. Την ε, περασμένη εβδομάδα επίσης υποβάλαμε κάποιες προτάσεις για τις διαρθρωτικές δράσεις και για την πολιτική συνοχή κατά την περίοδο κατόπιν του 2013. Αυτές οι προτάσεις περιέχουν πολλά στοιχεία απλούστευσης. Ενιαίο κανονισμό, κοινέ διατάξεις για όλα τα διορθωτικά ταμεία. Ανάπτυξη της Υπέδρου και το Ταμείο Ελίας. An important number of errors be Θα πρέπει να δούμε ότι αν εξορρονίσουμε τις κανόνες για τους δημόσιους διαγωνισμούς θα μειωθούν τα λάθη. Μια πράσινη βίβλος ε, έχει ήδη υποβληθεί και καλύπτει με ένα ευρύ φάσμα για την μεταρρύθμιση, την νομοθετική που θα γίνει και στόχος είναι το ότι τα χρήματα των συμβάσεων ε, πρόκειται να επενδύουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έχουμε τώρα την οικονομική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των κανόνων. Οπότε και για αυτόν τον τρόπο πρόκειται εμεί να εξετάσουμε πώς αυτές οι νέες ε, διατάξεις πρόκειται να βελτιωθούν στην πράξη την ενιαία αγορά είχαμε πει για αυτήν την νομοθετική πρόταση για το 2011. Οπότε και καλούμε τα άλλα κρατημέλη και τα, άλλα, δηλαδή τα κρατημέλη μάλλον και τα άλλα θεσμικά όργανα να θεωρήσει το ετήσιο πλαίσιο για να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση και επίσης τους μηχανισμούς διαχείρισης και ελέγχου για να είναι πιο αποτελεσματική και να εξασφαλιστεί ότι ο έλεγχος των δαπανών μας θα είναι αναλογικός, αποτελεσματικός και σωστή σχέση κόστους αποτελέσματος. Η τελευταία διαδικασία απαλλαγής ξεκαθάρισε ότι τα κράτη-μέλη θα να κάνουν περισσότερα για να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους και την κοινή διαχείριση. Έδειξε όμως ποια είναι τα όρια της Επιτροπής όσον αφορά το πόσο μπορεί να επηρεάσει, πόσο μπορεί να, να πει στα κράτη-μέλη όπως εδώ που θέλουμε να, τα κράτη-μέλη να αναφέρουν την καλύτερη διαχείριση για τους πόρους. Γι' αυτό και εμείς στο πακέτο συνοχής που ψήφισε την περσμένη εβδομάδα ε, βάλαμε και μία πρόταση που λέει ότι θα πρέπει να προχωρούμε σε καθαρή διόρθωση όταν έχουμε μία σειρά διορθώσεων στο σύστημα των κρατών μελών. Αυτό σημαίνει ότι όταν έχουμε κάποιου πόρου που περισσεύουν, τότε αυτοί δεν πάνε σε άλλο πρόγραμμα, αλλά επανέρχονται στον προπολογισμό ε, και συνυπολογίζονται ε, από το ποσό που γενικά παίρνει ένα κράτο μέλο. Κυρίε και κύριοι, σα εξήγησα ε, κάποιε συγκεκριμένε μα προτάσει, ούτω ώστε να δούμε τι βελτιώσει μπορεί να γίνουν. Και αυτόν τον τρόπο συμπληρώνουμε τι προσπάθειε που ήδη έχουν καταβληθεί τα τελευταία χρόνια και έτσι να έχουμε καλύτερη διαχείριση ήδη οι προσπαθειές μας έχουν αποδώσει καρπούς. Επίσης, απέδωσε η προσπάθεια μας για μείωση των λαθών. Πέρσι, το δικαστήριο είπε ότι το ποστό λάθος είναι μεταξύ 2 και 5% και ταυτόχρονα το δικαστήριο είπε για τις αιτήσει, ε, το δικαστήριο στο συνεδρικό συνέδριο είπε ότι το ίδιο ισχύει και για τις εκθέσεις. Ε, όλες. Τώρα προσπαθούμε να δούμε τι θα γίνει για την προϊόν προγραμματισμού, ούτως ώστε να έχουμε συγκεκριμένα μέτρα επί τη βάση της ε, απόφασης που θα ληφθεί με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο. Σας είπα τι έγινε με αυτά τα μέτρα, τι θα γίνει όταν αρχίσουν οι πραγματεύσεις με το Συμβούλιο με αυτές τις προτάσεις. Τώρα, δύο λόγια όσον αφορά την ετησία έκθεση για τις εσωτερικούς ελέγχους για τη χρήση 2010. Ε, αυτό το έγγραφο ήδη το έχετε λάβει και είμαι έτοιμος να το συζητήσουμε προσεχώς όταν Είναι Ενημερώνεται εδώ πέρα η αρχή επί της απολογής για το τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά το 2010, κάποιες συστάσεις και τη δράση που ανελήφθη επί τη βάση των συστάσεων. Και όλες οι συστάσεις ε, ε, ε όλες οι συστάσεις ήταν ε, αποδεκτές και αποφασίστηκε την ίδια χρονιά να ολοκληρωθούν αυτές οι ενέργειες που έπρεπε να γίνουν. Θεωρήθηκε ότι η IAS που υπάρχει εδώ και 10 χρόνια έχει φτάσει ικανοποιητικό επίπεδο οριμότητος. Οπότε και το στρατηγικό σχεδιασμό του IAS χαιρετίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς και οι ενέργειές της για εσωτερικό έλεγχο. Διακυβέρνηση, προτάσεις, τονίστηκε τι γίνεται όσον αφορά την πρόληψη της απάτης, την ανείχνευση αυτής και μας συνέστησαν να ενημερώσουμε, να επικαιροποιήσουμε τη στρατηγική μας. Να υπάρξει κάποιο, κάποιο σώμα που να ελέγχει την πολιτική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στρατηγικές ελέγχου. Είπαμε ότι εδώ υπάρχουν κάποια κενά. Η IIS είπε ότι θα πρέπει να υπάρξει προγραμματισμός για οικονομικούς ελέγχους πέραν του ενός έτους. Να δούμε τι γίνεται η διαδικασία ε, αποτίμησης των κινδύνων και να συντονιστούν μεταξύ τους οι υπηρεσίες. Οπότε είπαμε ότι έχουμε εδώ κάποιες προθεσμίες, το πρέπει να υπόψη κάποιες γενικές διευθύνσεις και ε, δεν, δεν τηρήθηκαν όμως πάντοτε αυτές που έταξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ότι έχουμε πρόγραμμα δράσης για τις ε, συστάσεις και οπότε και εμείς ε, εγκρίναμε τις προτάσεις αυτές για τα εγκάρσια ζητήματα όπως περιέχονται στις εκθέσεις και επίσης εκδώσαμε αυτή την ανακοίνωση κατά της απάτης που ευθυγραμμίζεται με τις προτάσεις του IAS. Οπότε γι' αυτό είπαμε ότι βελτιώντας τη στρατηγική θα έχουμε καλύτερη προστασία των ε, κοινοτικών οικονομικών συμφερόντων. Θα συμπληρωθούν διάφορες πρωτοβουλίες όπως η μεταρρύθμιση της, ε, της αντιμετώπισης της απάτης και της διαφθοράς. Όσον αφορά τώρα την καινούρια μας πολιτική για την πληροφορική. Ξεκίνησαμε μια καινούργια προσπάθεια το 2011 και έχουμε και δύο επιστολές που έχουμε συντάξει. Είμαστε βέβαιοι ότι έτσι θα έχουμε βελτίωση σε πολλά σημεία και πολλές οικονομίες. Προστίγες ελέγχου. Θέλουμε μια σειρά πρωτοβουλειών. Στοχευμένες, στοχευμένη Έλεγχη επιτόπου όσον αφορά την αναζήτηση αχρεωστήτων από κάποιους που έχουν λάβει χρήματα από τα διευθυντικά ταμεία με κατάλληλα συστήματα ελέγχου. Υπάρχουν τώρα τα προγράμματα δράσης και χρησιμοποιούνται εκεί που έχουν επισημανθεί μεγαλύτερη κίνδυνη. Τέλος, λάβουμε μια σειρά μέτρων για να βελτιωθούμε όσον αφορά την περιμερή για τις πληρωμές, αλλά και τους δικούς μηχανισμούς, ακριβώς όπως αναγνωρίζεται από τον Ευρωπαίο Διαδοσολαβητή. Όλα αυτά τα ζητήματα λήφθηκαν υπόψη για να, να δούμε τι θα κάνουμε για τις αδυναμίες, τι θα κάνουμε για τους κινδύνους που έχουν επισημανθεί. Και έτσι θα δούμε τι θα γίνει με αυτές τις συστάσεις που τώρα έχουν κλείσει 6 μήνες. Οπότε η Επιτροπή αυτού του ελέγχου υπενθυμίζει ποιε υπηρεσίε δεν έχουν κάνει αυτό το οποίο έπρεπε και ενημερώνεται ο Επίτροπος και όλο το Σώμα των Επιτρόπων. Εμείς με χαρά μας λέμε ότι υπάρχουν εξελίξεις συνεχώς θετικές για το γενικότερο επίπεδο αξιολόγησης. Ευχαριστώ και περιμένω πώς και πώς να τα συζητήσουμε. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Υπάρχει κάποιος ο οποίος θα ήθελε να κάνει ερωτήσεις εις ε, τον Επίτροπο σχετικά με την έκθεση. Ο εισηγητής μήπως θέλει να αναλάβει πρώτος τον ε, λόγο. Ε, επί του προκειμένου είμαι ο γυρεότερος στην Επιτροπή αυτή, ο πρεσβύτερ. Ε, αλλά ε, εγώ είμαι εισηγητής, λέει ο κ. Φέλνερ, οπότε... Καταρχήν θα ήθελα να προχωρήσω ένα επίπεδο πιο πέρα για να είμαι βέβαιος ότι κατάλαβα αυτά που έγραψε ο Επίτροπος και δεύτερον ε, για να μπορέσω να του κάνω και ερωτήσεις κατά τρόπον ώστε να ε, μπορεί αυτή η διαδικασία να έχει περισσότερη αξία για μας. Αλλά αυτό που βρήκα πιο ενδιαφέρον ήταν... το το κεφάλαιο σχετικά με, ε, τις, με τους εσωτερικούς ελέγχους αντιλαμβάνουμε ότι η πρώτη σχετική γνωμοδότηση ε, υποβλήθηκε το Μάιο εφέτος. Αντιλαμβάνουμε ότι αυτό είναι πολύ σοβαρό. Θα ήθελα όμως να ξέρω ποια είναι η προστιθέμενη αξία αυτής ε, της ε, γνωμοδοτήσεως για την γενική αξιολόγηση και τι καλύπτει. Δηλαδή, εάν φτάνει μέχρι και στους έλεγχο εντός των κρατών μελών ή σταματάει στα σύνορα σύνορα και αν ναι ποιο ήταν το νόημα και ποιο, ποια ήταν και η ετοιμιγορία αυτής της εκθέσεως διότι αυτό θα μας πει εάν είναι κάτι το οποίο θα συνεχίσει να ε, γίνεται και στο μέλλον. Μετά είδα δύο εκφράσεις Παραδείγματος χάρη, είδα ότι στον εσωτερικό έλεγχο στη σελίδα 4 η Επιτροπή θεωρεί ότι το 2010 κατατίστηκε μία μέθοδος διαδικαστική η οποία βοηθάει στην επίτευξη των οικονομικών στόχων εκτός από τους τομείς οικονομικής διαχείρισης όπου οι γενικοί διευθυντές είχαν επιφυλαχθεί σχετικά με την διαχείριση του κινδύνου στις σχετικές συναλλαγές. Όταν το διαβάζω όμως αυτό, αυτό που είναι ενδιαφέρον για μένα είναι τι σημαίνει αυτή η γνωμοδότηση διότι ε, αντιλαμβάνουμε ότι αυτό δεν είναι κάτι ε, δημόσιο άρα ε, αποκλειόμαστε και άρα θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η σημασία αυτών των παρατηρήσεων. διότι εδώ Μιλάμε ε, για την διαχείριση ε, του κινδύνου σε περιοχές όπου υπάρχει ε, κάποια αμφιβολία. Ποιο ήταν λοιπόν το αποτέλεσμα του οικονομικού ελέγχου. Εάν υπάρχει κίνδυνο στην οικονομική διαχείριση, εάν διατυπώθηκαν παρατηρήσεις, θα ήθελα να ξέρω ποιες ήταν αυτές οι παρατηρήσεις. Δεύτερον, Θέλω να προχωρήσω στο θέμα των επιφυλάξεων, διότι αντιλαμβάνομαι ότι παρόλο που πολύ σωστά η Επιτροπή λέγει ότι οι επιφυλάξεις από 20 μειώθηκαν σε 17 το 2010 ε, παρόλα αυτά επαναλαμβάνονται πολλές ε, δηλαδή 9 από τις 17 επαναλαμβάνονται αντιλαμβάνομαι ότι ο Επίτροπος Εμέτας είναι πολύ ευσυνείδητος προσπαθεί να βρει μία λύση και πρέπει να υπάρχει ανάληψη ευθυνών από τον κάθε επίτροπο. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω πόσο κατανέμεται ε, αυτή η ευθύνη μεταξύ των επιτρόπων για την εφαρμογή των προγραμμάτων για να μην υπάρχουν ε, ε, επαναλαμβανόμενες επιφυλάξεις διότι ίσως και οι οικονομικοί ελεγκτές είναι σε θέση να εκφραστούν επ' αυτού και ε, σχετικά με αριθμούς που προέκυψαν ε, σε διάφορες τομείς της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής να δουν ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη επί του θέματος. Προσπαθώ λοιπόν να ε, συγκρίνω τη συνθετική έκθεση με την παρουσίαση των ισολογισμών και είναι δύσκολο να την κατανοήσω διότι στη συνθετική έκθεση λέγεται ότι 97% από των συμπεφωνημένων διορθώσεων για τη συνοχή είχαν εφαρμοστεί μέχρι το τέλος του 2010 και μετά λέγεται ότι η εφαρμογή ε, για τις ε, οικονομικές ε, για τις οικονομικές προσαρμογές για την περίοδο 2006 με 2010 κάλυπταν μόνο το 58%. Άρα αυτά ε, είναι αντιφατικά. Από τη μία πλευρά μιλάμε για 97% και από την άλλη μεριά μιλάμε για 58%. Προσπαθώ λοιπόν να καταλάβω. Και τέλος, ε, το θέμα της συνοχής που είναι κάτι το οποίο θα ξανασυζητήσουμε ε, κατά την απαλλαγή αλλά στη σελίδα 19 λέγεται ότι για την πολιτική ε, συνοχής ε, τα λάθη εις την παρουσία στην αναφορά ήταν περισσότερα από ό,τι στο παρελθόν. Λοιπόν, θα ήθελα να μπορέσει η Επιτροπή να μας μιλήσει ε, ανοιχτά και να το συζητήσουμε με τους ε, το συζητήσουμε και με τον υπεύθυνο επίτροπο στη συνέχεια. Θα έρθει και αυτού η ώρα. Αλλά τώρα πολύ θα ήθελα να μας πει ο κύριος Σεμέτα γιατί είναι τόσο δύσκολο, παραδείγματο χάρη για τη Γενική Διεύθυνση Ρέτζιο, να μπορέσει να ισοσκελίσει τους λογαριασμούς της. Όπως είπα λοιπόν και στην αρχή, είναι σημαντικό να καταλάβει κανείς και να διαβάσει προσεκτικά το έγγραφο αυτό, διότι περιλαμβάνει πάρα πολλές ε, πληροφορίες και εφόσον πρόκειται και για μία συνθετική έκθεση και όπως άλλωστε ε, και ε, στην έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες είναι διοικητικές εκθέσεις είναι βασικό με να έχουμε την ερμηνεία από τους διαχειριστές αλλά καλό θα ήταν για μας συγχρόνως να έχουμε και κάποιον άλλον ο οποίος παρακολουθεί τα ίδια θέματα. Παραδείγματος χάρη το ελεκτικό συνέδριο, να έχουμε την άποψη του ελεκτικού συνεδρίου επ' αυτού. Δηλαδή αν όντως αντικατοπτρίζει ε, το έγγραφο αυτό την ε, κατάσταση των επιτευγμάτων ή προσπαθεί να αποκρύψει περισσότερα από ό,τι αποκαλύπτει. Θα πρέπει λοιπόν το ελεγκτικό συνέδριο να καταρτήσει μία δεύτερη γνώμη στην επόμενη ε, ανακοίνωση την οποία θα μας κάνει την επόμενη εβδομάδα. Ε, δυστυχώς ε, έχω ετοιμάσει ε, πολλές από τις σημειώσεις μου στα Σουηδικά. Αλλά εάν το ελεγκτικό συνέδριο μπορεί να περιλάβει τα στοιχεία αυτά στην ετήσια διαδικασία ή να παρουσιάσει ανεξαρτήτως την αξιολόγηση. Αν οι πληροφορίες είναι σωστές, εάν απαντούν τα ερωτήματα, εάν δεν αποκρύπτουν περισσότερα από ό,τι αποκαλύπτουν. Ελπίζω λοιπόν ότι με κατάλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί ίσως ε, δεν ήμουν πάντοτε πολύ σαφής. Θα... Σας ευχαριστώ πολύ. Να κάνω ένα μικρό σχόλιο. Να δώσω το λόγο καταρχήν στον κύριο Χατζημαρκάκη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, εκ μέρου μου, ε, σαν ε, προκάτοχος της εκθέσεω αυτή ε, από τον Κρίστοφελ Γέρνερ θέλω να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα ανοιχτά και ειλικρινά σχόλια, διότι βλέπουμε ότι πολλέ από τις απαιτήσει του Κοινοβουλίου πέρυσι έχουν ικανοποιηθεί. Αν δούμε δούμε πόσο περισσότερο έχουν κατακαιρματιστεί οι αριθμοί, πράγμα το οποίο οδήγησε σε μία αύξηση των κακών αριθμών για τα κράτη-μέλη, αλλά μου αποδειχνεί ότι όντως η Επιτροπή επεμβαίνει και γι' αυτό στο σημείο αυτό Κύριε Επίτροπε, θέλω να σας συγχαρώ, είναι ο σωστός δρόμος, πρέπει όμως έτσι να συνεχίσουμε, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι θα αντιμετωπίζετε αντίσταση από ορισμένα κράτη-μέλη. Θα ήθελα να ακούσω τη δικιά σας αξιολόγηση, αν με τα νέα μέσα τα οποία χρησιμοποιείτε ε, τα κράτη προσπαθούν να σας εμποδίσουν ή αν υπάρχει όντως μια επικοδομητική συνεργασία. Ε, καταρχήν λοιπόν όντως έχετε 2,7 ε, δισεκατομμύρια κατόπιν των αριθμών αυτών που δεν κατεβλήθηκαν και επίσης τα νέα συστήματα, ε, τα ε, συστήματα ελέγχου στα οποία είχε ζητήσει το Κοινοβούλιο τώρα έχουν εφαρμοστεί ε, ικανοποιητικά και αντιλαμβάνομαι ότι τα, στον τομέα της περιφερειακής πολιτικής 12 κράτη έχουν προβλήματα εφαρμογής ενώ στη Γεωργία μόνο τρίτη και συμφωνώ με τον Κρίστοφ Φέλνερ ότι η περιφερειακή πολιτική είναι ο πιο προβληματικός τομέας όπως ήταν και στο παρελθόν άρα πρέπει να κάνουμε κάτι ιδίω αν κοιτάξουμε τους αριθμούς στον τομέα συνοχής που είναι πέραν του 5% ενώ 5% των πληρωμών που αμφισβητούσε το ελεγκτικό συνέδριο και φαντάζομαι ότι αν το κοιτάξει κανείς από πιο κοντά ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί. Θα ήθελα λοιπόν ε, κατόπιν αυτού να συγχαρώ τον Πρόεδρο διότι βλέπω ότι υπάρχει μία αύξηση των κρατών οι ε, τα οποία υποβάλλουν μία σωστή δήλωση δηλαδή έχουν προσθεθεί η Δανία, η Ολλανδία, η Γερμανία και η Σουηδία και θεωρώ ότι αυτή η εξέλιξη είναι θετική. Μπορώ λοιπόν να ρωτήσω γιατί η συνθετική έκθεση αυτή δεν συνδυάστηκε με την έκθεση του εσωτερικού ελέγχου εφόσον όλοι οι συμμετέχοντες είναι εδώ. Γιατί δεν δόθηκε από κοινού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εφόσον η Επιτροπή, ε, το Κολέγιο των Επιτρόπων την απεδέχθη συγχρόνως ε, με την κεφαλαιοτική έκθεση και ε, ε, επεδόθη εις ε, τους ελεγκτές. Επίσης τι γίνεται με την ενημέρωση διότι είπαμε ότι πρέπει η Γενική Διεύθυνση να ενημερώνει καλύτερα τους τους ε, ε, επιτρόπους και να τονίζει ότι έχουν προχωρήσει αυτές οι συζητήσεις ε, γραπτός και επίσης όσον αφορά τον εσωτερικό έλεγχο θα ήθελα να μου πείτε τι νεότερα έχετε να μας ανακοινώσετε. Ευχαριστώ. Τώρα υπάρχει ακόμη ένας ομιλητής, ο κύριος Γκάιερ πρώτα. Με συγχωρείτε, εγώ δεν είμαι η κυρία που απουσιάζει. Ήμουνα εδώ και ήμουνα εδώ συνέχεια. Δεν έχω να προσθέσω πολλά σε αυτά που είπε ο και θα επανέλθω στο τέλος ε, της, ε, των σχολείων μου ότι δηλαδή ε, έχουμε μόνο μία περιορισμένη δήλωση αξιοπιστίας από το ελεγκτικό συνέδριο σχετικά με το 2010. Θα δούμε τι γίνεται στη συνέχεια αλλά δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι. Εγώ τουλάχιστον δεν είμαι και δεν επαρκούν αυτά για την εργασία εργασία της Επιτροπής αυτής. Ε, και με ανάμεικτα συναισθήματα διαπίστωσα ότι στον τομέα της συνοχής θα φτάσουμε στο 10% που δεν είναι ούτε βελτίωση ούτε επιδείνωση του ό,τι είχαμε δει πέρυσι και με ορισμένους συνεργάτες εις την σοσιαλδημοκρατική ομάδα εργασίας είχαμε την ε, ευκαιρία να ε, ακούσουμε τον Γενικό Διευθυντή για την Περιφερειακή ε, πολιτική ο οποίος μας είπε ε, τι προσπάθειες καταβάλει η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος για να μπορέσει να μειώσει αυτές ε, τις ε, αρνητικές αξιολογήσεις του ελεγκτικού συνεδρίου. Ο κύριος Σταυρακάκης και εγώ λοιπόν τον ρωτήσαμε αν είναι έτοιμος να έρθει στην Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού το οποίο να και την επόμενη φορά θα τον ακούσουμε διότι είναι η αχίλιος πτέρνα του ευρωπαϊκού προπολογισμού αυτό το θέμα και πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Αυτό που δεν με καθησυχάζει στο θέμα αυτό είναι ότι η δικιά του πρόγνωση ήταν ότι αν ακολουθήσουμε τις αυξομοιώσεις ε, ε, του, του επιχειρησιακού προγράμματος στα κράτη-μέλη δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει ότι το ποσοστό των σφαλμάτων θα αυξηθεί. Αυτός το έχει προεξοφλήσει, αλλά πολιτικά δεν μας καθησυχάζει καθόλου αυτό. Και τώρα έχω μία ειδική ερώτηση στον ε, Επίτροπο σε μέτα. Δεν είμαι βέβαιος εάν ο αριθμός των προγραμμάτων τα οποία έχουν διακοπεί στον τομέα της πολιτικής συνοχής ε, συνάδει με αυτό το ποσοστό των ε, σφαλμάτων ή όχι διότι ε, το, το γενικό πλαίσιο είναι ότι αν έχω προγράμματα τα οποία διακόπτω στα κράτη-μέλη λόγω σφαλμάτων και έχουμε ενθαρρύνει εις της, την Επιτροπή να το πράξει και τότε δεν εισραίει χρήμα στις χώρες αυτές και άρα δεν μπορούν να γίνουν και λάθη. Οπότε ε, αυτή η διακοπή της χρηματοδότησης έχει συνυπολογιστεί ε, στα, για τα προγράμματα που διακόπησαν ή όχι διότι τότε αυτό σημαίνει ότι μπορεί το ουσιαστικό ποσοστό να είναι πολύ υψηλότερο, στην οποία περίπτωση πρέπει να δούμε πώς το ποσοστό αυτό των ε, σφαλμάτων μπορεί να μειωθεί ε, γιατί η διακοπή των επιχειρησιακών προγραμμάτων είναι σοβαρό θέμα ιδίως όταν δεν έχουμε και πάρα πολλούς πόρους και είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να επηρεάσουμε τα κράτη-μέλη. Όσον αφορά την Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης ε, και Πολιτικής πολιτισμού και βλέπω 7,5% ποσοστό λάθους και ανικανοποιητικά έγγραφα, τότε νομίζω ότι στη διαδικασία απαλλαγής αυτό το θέμα είναι κάτι που πρέπει να δούμε πολύ συγκεκριμένα. Διότι αν κανείς δεν υποβάλλει επαρκή έγγραφα και δικαιολογητικά, αυτό σημαίνει πολλά. Δηλαδή, ε, εάν η η φωτοτυπία δεν είναι αναγνώσιμη, ο πάρεδρος στη δικιά μου περιοχή απορρίπτει το έγγραφο, το οποίο δεν σημαίνει ανεπαρκή ποιότητα, είναι ένα πρόβλημα τσαπατσουλιάς ε, και ε, δεν είναι επαρκής λόγος για να αρνηθούμε τη χρηματοδότηση, γι' αυτό και θα ήθελα να δούμε αυτό το πρόγραμμα δράσης και να δούμε πώς πρέπει να το προχωρήσουμε. Ολοκληρώνοντας πρέπει να πω ότι θα λάβουμε το πρώτο, την πρώτη έκθεση από το ελεγκτικό συνέδριο όπου θα έχουμε το σύστημα με τα πράσινα και κόκκινα σηματάκια δηλαδή να δούμε ε, πιο εμφανώς τι πήγε καλά και και όχι, αλλά στην πρώτη έκθεση απαλλαγής σε αυτήν την ε, θητεία είδαμε ότι το ποσοστό των σφαλμάτων ε, πρέπει να, να μειώνεται και αναρωτιέμαι αν ε, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι αξιόπιστη η παρουσίαση και φοβάμαι ότι το ίδιο θα συμβεί και σε αυτή την περίπτωση οπότε πρέπει να ε, καταλήξουμε στα πολιτικά συμπεράσματα. Η κυρία Κέσλερ Ευχαριστώ. Θέλω να κάνω δύο ερωτήσεις. Καταρχήν, το 2010 πιστεύαμε ότι πρώτη φορά θα ακούγαμε κάτι για τα νέα χρηματοδοτικά μέσα του προγράμματος μέχρι το 2013. Ποιες είναι τώρα οι εμπειρίες χρήσεως αυτών των μέσων και Πότε θα μας ενημερώσετε και επιπλέον η ε, έκθεση, η αναθεωρημένη ε, ανακεφαλωτική έκθεση ε, με οδηγεί να σκεφτώ ότι δεν πάμε καλά έτσι και είμαι βέβαιη ότι κάπου υπάρχει και, το, και η έκθεση των ελεγκτών την οποία δεν είχαμε σήμερα και πρέπει ε, να δούμε αν μπορούμε να ικανοποιηθούμε με την έκθεση αυτή διότι είχαμε ε, ζητήσει να υπάρχει πάντοτε η έκθεση του εσωτερικού ελέγχου μαζί με την ανακεφαλωτική. Κυρία Αντρέασεν. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Η πρώτη ερώτηση που εγώ θέλω να υποβάλω στον κύριο της Επιτροπής είναι γιατί αποφάσισε να καλέσει αυτό το σύνολο των επιφυλάξεων μιας, ως μια σύνδεση επιτευμάτων της Κομισιόν, γιατί εγώ δεν θεωρώ πως είναι επιτεύγματα αυτά καθόλου. Ε, Μάλιστα, αντιθέτω, το ελεγκτικό συνέδριο εξακολουθεί να επιμένει για το υψηλό επίπεδο σφαλμάτων ε, και εξακολουθεί αυτό να υπάρχει και στι παρατηρήσει του Γενικού Γραμματέα. Αν μιλά για την μείωση από το 20 στι 17 επιφυλάξει, πραγματικά είναι πολύ σφαλμένο αυτό, γιατί το 2009 ε, υπήρχαν 16 επιφυλάξεις και το 2007 17 και το 2006 20, δηλαδή ανεβοκατεβαίνουμε. Αυτό συμβαίνει και αυτό προκύπτει και από το ελεγκτικό συνέδριο για την έκθεσή του. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν πού βλέπει τα επιτεύγματα. Επίσης ανέφερε ε, ποιες είναι οι προτάσεις για βελτίωση και είναι πραγματικά οι ίδιες που έχουν ανεφερε ποιε ειναι οι εδώ και δύο χρόνια τουλάχιστον και παραπάνω η καταποκοπή ποσά, η χρήση των συστημάτων εποπτείας και ελέγχου και νομίζω πως σε αυτή τη φάση θα έπρεπε να βλέπουμε τα αποτελέσματα αυτών των βελτιώσεων. Ενώ δεν υπάρχουν πραγματικά αποτελέσματα. Θα ήθελα επίσης να ρωτήσω τον κύριο Σεμέτα για αυτό το πίνακα που έχουμε στη σελίδα 16 όπου δείχνει τις εξαιρέσεις, τα ποσά δηλαδή ανάκτησης που έχουν ε, αρθεί. Και θα, θα ήθελα να γνωρίζω για ποιον λόγο έχουν ε, δοθεί αυτές οι εξαιρέσεις. Επίσης, θα ήθελα να γνωρίζω ποιες είναι οι χώρες στις οποίες θα μπορούσε να υπάρξει δήλωση εξοπιστίας. Βλέπω τη Γερμανία, αλλά η Γερμανία αναφέρεται στο Ταμείο Συνοχής ως ένα από τα κρατη όπου υπάρχει ένα ψηλός βαθμός αντικανονικότητας. Υπάρχει εξήγηση γι' αυτό και πώς αυτό ταιριάζει με τη δήλωση της Γερμανίας. Σας ευχαριστώ. Τον λόγο έχει η κυρία Ιβανόβα. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για την παρουσίασή του. Εγώ δεν έχω πάρα πολύ να πω γιατί τις περισσότερες ερωτήσεις έθεσαν ήδη συνάδελφοι. Απλώς θα ήθελα να πω πως καλωσορίζω τις πληροφορίες που μας δόθηκαν για την αποτελεσματικότητα των ελεκτικών συστημάτων στα διάφορα κράτη-μέλη. Επιμείναμε γι' αυτό στην προηγούμενη απαλλαγή και νομίζω πως είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ποιο σύστημα ελέγχου ήταν επαρκές και ποιο όχι ώστε να μπορούμε να δώσουμε σωστές συνταγές. Ε, ωστόσο θα ήθελα να ζητήσω από τον Επίτροπο να διευκρινίσει κάπως περισσότερο ποια ήταν η πρόοδος που σημειώθηκε στη βελτίωση το, γενικότερα των μηχανισμών ελέγχου. Ξέρω πως ανέφερε πλέον ε, στόχους ελέγχου, αλλά μήπως θα μπορούσε να μας δώσει λίγες περισσότερες πληροφορίες για την πρόοδο που σημειώθηκε. Thank no Σας ευχαριστώ, δεν βλέπω άλλους να ζητούν το λόγο, οπότε θα ήθελα να ρωτήσω το ελεγκτικό συνέδριο ποια άποψη έχουν ε, για την πρόταση του εισηγητή το συνέδριο να δώσει ένα σχόλιο για την ε, συνοπτική έκθεση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Φυσικά και συμμεριζόμαστε την ανησυχία του εισηγητή σας όσον αφορά τη σκοπιμότητα ε, δημιουργίας μιας, μάλλον ύπαρξης μιας εξωτερικής ε, εκτίμησης ή κρίσης ε, της ε, Κομισιόν για την ίδια της τη δραστηριότητα. Μάλιστα, έχουμε τέτοια εξωτερική, μάλλον μας παρέχουμε αυτή την εξωτερική γνωμοδότηση για στο τέλος κάθε κεφαλαίου της ετήσιου συνεδρίου υπάρχει ένα τμήμα το οποίο είναι αφιερωμένο στην ανάλυση της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων κάθε γενικής διεύθυνσης. και πολύ συχνά οι κρίσεις του συνεδρίου ε, διαφέρουν από τις κρίσεις της ίδιας της Γενικής Διεύθυνσης για την ίδια της τη δραστηριότητα. Τώρα, το νέο χαρακτηριστικό περί του οποίου μιλάμε είναι η συνθετική αυτή συνοπτική έκθεση που από τη φύση της παρουσιάζει μια σύνθεση, μια σύνοψη των λεπτομερών πληροφοριών που παρέχονται στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της κάθε γάμα δέλτα. Πέρυσι το συνέδριο νομίζω ήταν για πρώτη φορά είδε τη συνθετική έκθεση. Δημοσιεύσαμε ένα σύντομο σχόλιο για την έκθεση αυτή τη συνοπτική. Φέτος ολοκληρώνουμε την ετήσια μας έκθεση που θα δημοσιευθεί τον Νοέμβριο και στην έκθεση αυτή θα υπάρξει ένα κομμάτι που θα είναι αφιερωμένο στην ε, ε, συνοπτική έκθεση. Και Πάλι θα ήθελα να επαναλάβω ότι η πραγματική λεπτομερής κρίση του συνεδρίου Έγινε στην κρίση που κάνει για κάθε ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων κάθε γάμα δέλτα. Γιατί σε αυτό το επίπεδο λεπτομέρειας μπορούμε εμείς να προβούμε σε έλογα σχόλια για τις, ε, τα επιτέματα της κάθε γάμα δέλτα. Αλλά επίσης σχολιάζουμε και την συνοπτική παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων. Ευχαριστώ. Ε, εμείς ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Μάλιστα. Ο εσωτερικό ελεγκτή, ο κύριο Γκρέι, θέλει να σχολιάσει κάτι ή το αφήνετε τον ε, επίτροπο. In that case you have the floor. Happy to come. Ε, εσύ γιατί το λόγο. Ναι, ευχαρίστω να σχολιάσω, αλλά ίσω καλύτερα είναι να τα πει ο επίτροπο. Μάλιστα. Το λόγο έχει ο επίτροπο τότε. Chairman, if you would agree, I will start and then... Αν συμφωνείτε, Πρόεδρε, θα ξεκινήσω εγώ και ο εσωτερικό ελεγκτή να απαντήσει στα σχόλια που συνδέονται άμεσα με τη δική του δραστηριότητα. Καταρχήν σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις και για το ότι θίξατε τόσα θέματα. Θα ξεκινήσω με τις παρατηρήσεις του εισηγητή. Καταρχήν όσον αφορά την γενική άποψη. Θα πρέπει να σας πω, ήταν πρώτη φορά στην Επιτροπή όπου η εσωτερική, ο εσωτερικός μας έλεγχος εκπώνησε γενική έκθεση και δεν γνωρίζω κανένα άλλο δημόσιο θεσμικό όργανο τουλάχιστον στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου να γίνεται τέτοιου είδους έκθεση ε, από τον εσωτερικό ελεγκτή σε τόσο περίπλοκο μάλιστα θεσμικό όργανο. Νομίζω πως είναι λοιπόν πολύτιμο αυτή η προσπάθεια γιατί η γενική προετοιμασία για αυτή την γνωμοδότηση απέτησε έντονη συνεργασία ανάμεσα στην υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου και τις ε, εσωτερικές δυνατότητες ελέγχου σε κάθε γαμαδέλτα. Γι' αυτό οδήγησε σε πολύ καλύτερη κατανόηση για τις κατάστασεις στις διάφορες γάμα δέλτα. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στον Brian Gray για να σας εξηγήσει το πεδίο ε, που καλύπτει η γνωμοδότηση και επίσης το νόημα των παρατηρήσεών του. Να σας πω ότι Συζητήσαμε την έκθεση αυτή στην ε, Επιτροπή Προόδου του Οικονομικού Ελέγχου, ε, όπου συμμετέχουν 7 επίτροποι, αλλά και εξωτερικά μέλη και αναγνωρίστηκε η προστεθέμενη αξία της εν λόγω έκθεσης και επιβεβαιώθηκε η ανάγκη για συνέχιση αυτής της εργασίας. Σε σχέση τώρα με τις επιφυλάξεις. Τις επαναλαμβανόμενες επιφυλάξεις. θα πρέπει να σας πω πως έχουμε γενικά διαδικασίες που απαιτούν κάθε επίτροπος να συζητά με την ε, υπηρεσία του και να ελέγχει τις υπηρεσίες του τουλάχιστον δύο φορές ετησίως. Και φυσικά το θέμα της επιφύλαξης είναι κάθε φορά το θέμα κλειδί σε αυτού του είδος της συζητήσεις. Από την άλλη πλευρά, επίσης αποφασίσαμε να τονίσουμε πολύ περισσότερο αυτά τα θέματα μέσα στο πλαίσιο της Επιτροπής Προόδου του Οικονομικού Ελέγχου, του Εσωτερικού Οικονομικού Ελέγχου. Και κάθε φορά που προκύπτει ένα θέμα σε κάποια γενική διάθεση, παρακολουθούμε την εξέλιξη μέσα από αυτήν την Επιτροπή εσωτερικού οικονομικού ελέγχου και προόδου αυτού. Έπειτα έχουμε την εφαρμογή και την παρακολούθηση της ανάκτησης. Η διαφορά στους λογαριασμούς ε, στην ε, συνθετική έκθεση μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι έχουμε ε, στοιχεία που εφαρμόζονται σε επίπεδο που εκτελούνται σε επίπεδο κράτους μέλους, ενώ στο Συμβούλιο έχουμε τον ε, υπεύθυνο λογιστικού ελέγχου που αναφέρει τα στοιχεία. Ίσως αυτό να οφείλεται. Έχουμε στους λογαριασμούς ανακτήσεις που έχουν εγκριθεί από τον ε, υπεύθυνο. Και έπειτα Όσον αφορά την προστιθέμενη αξία της ε, συνοπτικής έκθεσης, φυσικά αυτή είναι μια έκθεση που συνοψίζει τα συμπεράσματα που έχουν προκύψει τόσο σε επίπεδο ετήσιας δραστηριότητας και των σχετικών εκθέσεων, καθώς και των συστάσεων που έχουν υποβληθεί από την Γενική Υπηρεσία Οικονομικού Ελέγχου. Αυτή είναι μια ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων για την συνοχή. Θα ήθελα να σας καλέσω μάλιστα να την μελετήσετε. Και αυτό θα απαντήσει και σε πολλές ερωτήσεις που ε, τέθησαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το ποια συγκεκριμένα μέτρα εφαρμόζονται όταν ο Γενικός ε, Διευθυντής εκφράζει επιφυλάξεις και ο κύριος Χαζημαρκάκης τον έφερε στην παρέμβασή του σε σχέση με τον αυξημένο αριθμό των κρατών μελών που είναι αντικείμενο επιφυλάξεων από τον Γενικό Διευθυντή. Εδώ πρέπει νομίζω να σκεφτούμε πώς θα γίνουν βελτιώσεις σε επίπεδο κρατών μελών. Γιατί όταν μιλάμε για το επίπεδο σφαλμάτων, η μεγαλύτερη πλειοψηφία τους ε, συγκεντρώνεται στην κοινή διαχείριση και σε επίπεδο κρατών μελών. Ο κύριος Χατζημαρκάκης επίτης ρώτησε για την αντίδραση των κρατών μελών στην αυξημένη διακοπή πληρωμών. Θα πρέπει να σας πω το 2010 διακόψαμε 49 πληρωμές για το Ταμείο Συνοχή, 12 πληρωμές για το Κοινωνικό Ταμείο καθώς επίσης και εφαρμόσαμε την ακύρωση, την αναστολή μάλλον, ε, έξι πληρωμών. Είναι ένα μέσο το οποίο μας επιτρέπει να βελτιώσουμε τη διαχείριση και τα συστήματα ελέγχου των κρατών μελών. Διότι η διακοπή δεν σημαίνει απλά ότι διακόπτουμε την πληρωμή και περιμένουμε και βλέπουμε, αλλά όταν διακόπτουμε την πληρωμή ζητάμε από το κράτος μέλος να προβεί σε συγκεκριμένε ενέργειες ώστε να διορθώσει την κατάσταση και την ε, διαχείριση και το σύστημα ελέγχου και μόνο όταν έχει γίνει αυτό από το κράτος μέλος, τότε μόνο μπορεί να συνεχιστεί οι πληρωμές. Είναι ένα πολύ ε, δυνατό μέσο λοιπόν που έχουμε στη διάθεσή μας. Φυσικά δεν αρέσει και πολύ στα κράτη-μέλη γιατί διακοπές προγραμμάτων μπορεί να σημαίνουν τεράστια ποσά και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την κατάσταση της λιτότητας. Δεν είναι πολύ ευχαριστημένα όλα τα κρατημέλη με αυτή την κατάσταση, αλλά εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να γίνεται αυτή η διαδικασία και, και μια νέα πρόταση για τα Ταμεία Συνοχής προτείνει την παράταση της περίοδου διακοπής από τους 6 στους 9 μήνες για να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα μέσα ακόμα πιο αποτελεσματικά. Σε σχέση λοιπόν με την έκθεση τη συνοπτική και την ε, έκθεση εσωτερικού ελέγχου, οικονομικού ελέγχου, Πιστεύω πως πρόσφατα σας δόθηκε η εκθέση σύμφωνα με το άρθρο 86.4 όπου ο ιστορικός ε, ε, ελεγκτής ελέγχει το τι έχει γίνει σε επίπεδο ιστορικού οικονομικού ελέγχου και αυτή η έκθεση είναι αντικείμενο συζήτησης εδώ στο Κοινοβούλιο και ίσως αυτό που έχετε υπόψη είναι αυτή η γενική έκθεση που εκπώνησε ο εσωτερικό ελεγκτή, ο Μπρέν λοιπόν να με βοηθήσει για να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα. Αλλά το θέμα πάντω είναι ότι είναι μια γενική γνώμη, η γνωμοδότηση για τη διαχείριση και φυσικά υπάρχει ανάγκη να αξιολογήσουμε ποιες θα ήταν οι συνέπειες αν αυτή η συνολική εσωτερική γνωμοδότηση δημοσιευθεί και μήπως θα πρέπει πρώτα, μήπως αυτό θα μείωνε την προστιθέμενη αξία αυτής της έκθεσης. Και αυτό είναι ένα θέμα στο οποίο ίσως ο Brian Gray θα μπορούσε να επεκταθεί κάπως περισσότερο. Τώρα, σε σχέση με τη διαφορά στα σφάλματα αυτό που ανέφερε ο κύριος Γκρέι, είναι αλήθεια ότι τα ασφάλματα διαφέρουν μεταξύ τους. Θα πρέπει αυτό να το εξετάσουμε πιο σοβαρά, αλλά φυσικά το ελεγκτικό συνέδριο αναγνωρίζει μόνο τα ασφάλματα εκεί όπου υπάρχει σημαντική επιρροή αυτών σε σχέση με την αποτελεσματικότητα των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου. Ε, πολλά από τα σφάλματα συμβαίνουν στο πρώτο επίπεδο ελέγχου, δηλαδή στο επίπεδο ενδιάμεσων οργανισμών όπου δεν γίνονται όλοι οι έλεγχοι με τον σωστό τρόπο. Και τώρα εξετάζουμε το πώς θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση στο πρώτο επίπεδο ελέγχου, διότι αν σε αυτό το επίπεδο μπορέσουμε να μειώσουμε τα σφάλματα, Αυτό θα οδηγήσει σε βελτίωση της κατάστασης γενικότερα στην ε, πολιτική συνοχής. Uh, uh, Η κυρία Γκρέσλε μίλησε για το θέμα της έκθεσης εσωτερικού οικονομικού ελέγχου και τη συνοπτική έκθεση και νομίζω ότι σε αυτά θα επεκταθεί περισσότερο ο Μπράιαν. Και όσον αφορά την χρήση των ε, δημοσιονομικών μέσων, ελέγχθηκαν και αναλύθηκαν κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και του ελέγχου των λογαριασμών της Επιτροπής ο αρμόδιος ε, του λογιστικού ελέγχου πρόσεξε ιδιαίτερα αυτό το ζήτημα γιατί τα χρηματοδοτικά μέσα αναγνωρίζονται ως ε, πληρωμές. Έχει γίνει τεράστια δουλειά πάνω σε αυτό. Θα μπορούσε να εξηγήσει με περισσότερες λεπτομέρειες αυτό το θέμα. Σε σχέση με την ερώτηση της κυρίας Αντρέασεν για τις εξαιρέσεις, Είναι απέτηση σύμφωνα με τους ε, κανόνες ε, του ε, δημοσιονομικού μας κανονισμού να ζητώνται εξαιρέσεις για την Κομισιόν και εξηγείται ως εξής. Γίνεται αυτό όταν η νομική υπηρεσία αναγνωρίζει πως δεν υπάρχει δυνατότητα για ανάκτηση των ποσών λόγω νομικών περιορισμών. Αυτή είναι η εξήγηση αυτού του πίνακα στην ε, συνοπτική έκθεση. Και κάθε ένα από τα νούμερα που έχετε στη συνοπτική έκθεση θα εξηγηθεί από τις συγκεκριμένες νομικές διατάξεις που δεν επιτρέπουν να γίνει η ανάκτηση των ποσών αυτών. Μάλλον εκάλυψα τις ερωτήσεις της κυρίας Ιβανόβα σε σχέση με διαχείριση και έλεγχο και τη σχετική δελτίωση που θέλουμε να επιφέρουμε ε, ε, μέσω των ερωτήσεων και απαντήσεων των άλλων ε, βουλευτών. Άρα, απλώς θα περιοριστώ να σας πω ότι... Όσον αφορά το νέο πρόγραμμα, εμείς σαφώς θα προβούμε σε διατύπωση προτάσεων νέων μέτρων. Αυτά τα οποία προανέφερα θεωρώ ότι το ζήτημα της καθαρής διόρθωσης είναι νέα έννοια όσον αφορά την διαχείριση των διορθωτικών, συγγνώμη, του, το, των ταμείων συνοχής. Εάν εγκριθεί από Συμβούλιο και Κοινοβούλιο, αυτό στην πράξη θα σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη δεν θα είναι εις θέση να επαναχρησιμοποιήσουν πόρους που επρόκειτο να διατεθούν εις μη επιλεγέντα προγράμματα ε, τα οποία περίφθησαν λόγω παραβίασης των κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις και διαγωνισμούς. το οποίο φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι τότε είναι θέμα της διάθεση πόρων γενετικών προς το κράτο μέλο συνολικά, γενικά. Πάντως, εδώ έχουμε και άλλα στοιχεία σε αυτή την πρόταση. Έγινε έγκριση της προτάσεω την περασμένη εβδομάδα. Θα δείτε επομένω ε, όλες τις διαστάσεις και παρακαλώ προσέξτε τα θέματα της απλούστευσης των διατάξεων αλλά και τα του δημοκρατικού ελέγχου, της λογοδοσίας όπως λέμε, των κρατών μελών για τα συγκεκριμένα μέτρα τα οποία προτείνονται σε αυτό το έγγραφο. Και τώρα, δώσουμε τώρα το λόγο τον Μπράιαν και στον Φιλίπ για να διευκρινίσουν τα θέματα αυτά. Okay, Mr. Gray, you have the floor. Uh, thank you, Mr. Gray, έχετε το λόγο τώρα για να απαντήσω στις ερωτήσεις του κ. Φιέρνερ ε, ποια είναι η γενική μου απάντηση σχετικά με την προστιθέμενη αξία. Ε, νομίζω το σύστημα αυτό υπάρχει εδώ και 10 χρόνια και στα 10 χρόνια κάναμε ορισμένους οικονομικούς ελέγχους και πιστεύω ότι μετά από 10 χρόνια έπρεπε ε, πλέον να εξασφαλίσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να την καθησυχάσουμε ότι το, ο έλεγχος αναφέρεται σε όλα τα συστήματα που έχουν σχέση με την οικονομική διαχείριση στην Ευρώπη. Έχουμε λοιπόν κάνει τα τελευταία τρία χρόνια προσαρμογές στα προγράμματά μας και μπορούμε να παράσχουμε αυτή τη διαβεβαίωση. Ιδίως όσον αφορά τον τομέα των δαπανών και ουσιαστικά η προστιθέμενη αξία είναι ότι όχι μόνο κοιτάξαμε τα στοιχεία αλλά ότι εξετάσαμε και πώς προχωράνε όσον αφορά την οικονομική διαχείριση αλλά και τη μη οικονομική διαχείριση το θέμα του τρόπου με τους οποίους της διαφανείας και του, της ηθικής πτυχής του συστήματος νομίζω ότι είμαστε ικανοποιημένοι. Είμαστε εσωτερικοί ελεγκτές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σταματάμε δηλαδή στην πόρτα της Επιτροπής. Ενώ η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή του προϋπολογισμού ακόμη και αν είναι έμεση η εφαρμογή αυτή ή εξωτερική. Οπότε πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι και αυτές οι κινήσεις γίνονται σωστά και αν πρόκειται ε, για εφαρμογή την οποία μοιράζεται με τα κράτη-μέλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την ευθύνη να εφαρμόσει ε, τις ε, λογιστικές μεθόδους και το πράτη για να αξιολογήσει τους ελέγχους και να αποφασίσει βάση αυτών εάν χρειάζονται διορθώσεις ή διακοπές της χρηματοδότησης και αυτό έχει γίνει. Βλέπουμε λοιπόν πώς αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πρόβλημα αυτό, τι κάνει και προσέχουμε πάρα πολύ τις γενικές διευθύνσεις συνοχής αλλά και γεωργίας για να είμαστε βέβαιοι ότι εφαρμόζουν σωστά τις διαδικασίες και τις ε, λογιστικές μεθόδους όσον αφορά τη διακυβέρνηση ε, και την εφαρμογή της. Πρέπει να καταρτήσουμε ε, προδιαγραφές και αυτός είναι ο στόχος μας. Να εξετάζουμε τους ελέγχους σε όλα τα επίπεδα ε, και όλες τις διαδικασίες. Έχουμε δηλαδή διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου οι οποίες προσαρμόζονται στις εθνικές προδιαγραφές όταν εξετάζουν αυτό το χρόνο. Τελικά βέβαια τίποτα δεν είναι τέλειο. Έχουμε συνεργαστεί με τους ε, γενικούς διευθυντές, έχουμε κάνει πολλές ε, διμερείς ε, συναντήσεις για να συμφωνήσουμε τις επιφυλάξεις. Δηλαδή πού θα αναφέρονται επιφυλάξεις στην ετήσια έκθεση του Γενικού Διευθυντή. Ε, και συμφωνήσαμε ότι οι επιφυλάξεις του εσωτερικού ελεγκτή της Επιτροπής βασίζονται στην σωστή ε, διαδικασία εσωτερικού ελέγχου. Αναφερθήκατε στις επιφυλάξεις που επαναλαμβάνονται, είτε διότι παραμένει κανείς πάνω από το 2%, οπότε κοιτάμε ε, αν η έρευνα κάνει αυτά τα οποία πρέπει και να εξασφαλίσουμε ότι σε κάθε τομέα υπάρχει η σωστή δομή ελέγχου και ότι αναλαμβάνονται τα διορθωτικά μέτρα τα οποία επιβάλλονται. Είδατε ότι είπαμε ε, ότι ορισμένες ε, ε, επιφυλάξεις παραμένουν οι ίδιες ή επαναλαμβάνονται επιφυλάξεις οι οποίες όμως αναφέρονται σε διαφορετικά θέματα διότι έχουν αναλυφθεί διορθωτικές ενέργειες. Θέλω επίσης να σας πω ότι δεν καλύψαμε το Γαλιλαίο, καλύψαμε τα πάντα πλην του Γαλιλαίου, δεν έχουμε τελειώσει εκεί ε, τον ε, έλεγχο και γι' αυτό το πρόγραμμα αυτό θα περιληφθεί ε, στο, την έκθεση εσωτερικού ελέγχου εφέτος και είδαμε ότι και εκεί πρέπει να γίνει ακόμη δουλειά για να εφαρμόσουμε τις επιταγές του ελεκτικού συνεδρίου να βελτιώσουμε το επίπεδο όσον αφορά τις δευτέρου βαθμού ε, συναλλαγές όπου δεν έχουμε σαφή εικόνα του τρόπου διεξαγωγής και επίσης πρέπει να υπάρχει ε, ένας ε, καλύτερος συντονισμός των ελέγχων των εμπλεκομένων ε, γενικών διευθύνσεων <clears throat> και να μην περιμένει κανείς τις εντολές του ελεκτικού συνεδρίου αλλά να κάνει σωστά τη δουλειά του. Αυτό θεωρούμε ότι είναι πολύ βασικό και τα έχουμε γράψει πολύ πιο λεπτομερό. Τώρα για το εάν πρέπει να δημοσιευθεί ή όχι. Εμείς ε, τις 86 εκθέσεις μας τις υποβάλλουμε στα θεσμικά όργανα και μετά συνοψίζονται σε μια συνθετική έκθεση. Και η συνθετική αυτή έκθεση ε, απεικονίζει σωστά και συνοψίζει την θέση μας στις πρώτες σελίδες. Σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Thank you, Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα-πρώτα για την ερώτηση του εισηγητού. Υπάρχει προοπτική Υπάρχει μια άποψη τέλο πάντων και το διαχείριση και δεν υποφορά την λογιστική, το 75% αυτό εκτελούνται, υπορροφούνται γιατί αυτό έχει γίνει ω ε, διόρθωση, γιατί αυτό έχει αφαιρεθεί από το κόστο. Όμω έχουμε κάποιε τέτοιε δηλώσει που βρίσκονται στην φάση του κλεισίματο και τώρα τι ε, ελέγχουμε από το ε, γραφείο έγκριση και δεν πρόκειται να εξομπούν στου λογαριασμού προ το παρόν. Επομένω, εάν θέλετε να δείτε τι κάνουν τα κράτη-μέλη, ε, έχουν πάει στα κατημέρια αυτά τα χρήματα αλλά δεν βρίσκονται στους λογαριασμούς γιατί όλη αυτή η δήλωση ακόμα δεν έχει εγκριθεί από τον ε, ε, ε το 632 5-6 ξεκάθαρες γραμμούλες πάλι πολύ βασικό είναι λοιπόν κάτι το οποίο ακόμα δεν έχει ε, ο, ο, ο αδειοδοτών τέλο δεν το έχει εγκρίνει τώρα για την κυρία Γκρέσλη Εάν κατάλαβα το οποίο ρωτήσατε καλά κύριε Γκρέσλε, αυτό αφορά το κατά πόσον το μέσο χρηματοδότησης αποδίδει για τον Επίτροπο Τώρα έχουμε αυτή την βασική διόρθωση για αυτού του προσωρινού λογαριασμού όσον αφορά αυτά τα μέσα χρηματοδότηση για του προσωρινού λογαριασμού του 2000. Οπότε αυτά τα έχουμε ολοκληρώσει διότι διαπιστώσαμε ότι κατά, τη, κατά το, την ολοκλήρωση του ελέγχου των λογαριασμών και θα πρέπει σε αυτό να είμαι πάρα πολύ ειλικρινή, όπω διαπιστώθηκε από το Ελληνικό Συνέδριο κατά το δικό του το έλεγχο ότι βρήκαν αυτό που βρήκαν και κατόπιν είπαν ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να δώσουν ενδελεχή ενημέρωση όσον αφορά αυτά τα ποσά ε, που προέρχονται από τους καταβάλλοντες οργανισμούς που δεν πάνε στους ε, ευεργετούμενους αλλά πάνε στους δικαιούς αλλά πρόκειται για κάποια μεταφορά πόρων για διάφορους λόγους όμως για διάφορους λόγους αυτά δεν έχουν προωθηθεί άμεσα επομένως θα πρέπει να ε, ξαναμπεί στον ισολογισμό το το ποσό. Μην σας πω τώρα τις λεπτομέρειες. Όλα αυτά έχουν τακτοποιηθεί, όλα έχουν διορθωθεί και έχουν ε, ικανοποίησει τον ελληνικών συνέδρων. Να μην σας πω τώρα τη, γνώμη τους, αλλά από δική μας πλευρά, από πλευράς ε, λογιστικής, έχουμε αυτή τη σημείωση 252 μπορεί να βρείτε αυτά τα στοιχεία. Όμως το πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα νομίζω ότι το 2011, θα, θα πάει και το 2010 και πριν το 2010 δεν το τίποτα. Επομένω, παρόλα αυτά είμαστε ακόμα σε φάση του ρονταρίσματος και αν θέλετε μπορείτε να υποβάλλετε και άλλες ερωτήσεις για τους ε, συναδέλφους. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Πριν δώσουμε τώρα το λόγο στον εισηγητή να συνοψίσει, υπάρχει κάποιος άλλος από τους συναδέλφους που θέλει κάτι άλλο να πει. Κύριε Γκρέσλε. Ευχαριστώ. Ε, αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με τα οικονομικά μέσα ή στα διαρθρωτικά τη, ταμεία άνοιξαν μία τράπεζα μένα αλλά δεν μοίρασαν τα, τους πόρους απλώς τους διατηρήσαμε. Ρώτησα λοιπόν αν κατάλαβα καλά ότι αυτοί οι οποίοι χρηματοδοτήθηκαν από τα χρηματοδοτικά μέσα κράτησαν τα χρήματα και δεν τα μεταβίβασαν. Και αυτό με απασχολεί και πάλι με τον δημοσιονομικό κανονισμό διότι ε, θα πρέπει να δεχθούμε σημαντικές τροπολογίες στα θέματα αυτά. Πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι ξέρουμε περισσότερα για τον final beneficiary και για το ποσό. Τρίτον, ε, όντως έτσι είναι ότι όλο το ποσό πληρώνεται σε μία φορά στα δημοσιονομικά μέσα ε, ε, ή αν αυτά διαρκούν 20 χρόνια πληρώνεται μόνο μία δόση. Αυτή είναι λεπτές ισορροπίες σε αυτό το τομέα διότι αν έχει κάποιος τα χρήματα αυτά και εργάζεται μαζί τους θα ήθελα να μου διευκρινίσετε πώς ακριβώς γίνεται. Ο κύριος Οντί. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τη στιγμή όπου ξεκινάμε ε, την ε, κοινοβουλευτική διαδικασία της απαλλαγής η συνθήκη προβλέπει ότι το Κοινοβούλιο για να μπορέσει να αποδώσει την ε, θέση του πρέπει να έχει μία βεβαίωση εξασφάλισης διασφάλισης η οποία να αναφέρεται και στους λογαριασμούς και στην αξιοπιστία των ε, ε, ε, ενεργειών στις οποίες αναφέρεται. Λοιπόν, ναι μεν έχουμε μία θετική γνωμοδότηση για, το, για τους ε, λογαριασμούς και για την ε, ε, δήλωση, δήλωση για τους λογαριασμούς αλλά δεν ξέρω αν μέχρι τις 10 Νοεμβρίου θα έχουμε όλα τα αναγκαία έγγραφα σχετικά με τους λογαριασμούς αλλά και με τις υποκείμενες εργασίες διότι το 2000 2009 ε, ε, δεν είχαμε πλήρες έτος, το έχουμε όμως τώρα. Και άρα το ελεγκτικό συνέδριο σκέφτεται πόσο θα συντάξει αυτή την έκθεση για τον εσωτερικό έλεγχο όπως μας ε, υπέδειξαν οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ. Μπορεί να σχολιάσει το δικαστήριο. Ναι, ναι, βεβαίως κύριε Πρόεδρε. Για να πούμε κάτι. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Όχι. Είναι κάπως περίπλοκο, αλλά αυτό κατά κάποιο τρόπο επαιδεί και η συνθήκη. Έχουμε δύο είδη γνωμοδοτήσεων. Μία όσον αφορά τους λογαριασμούς και ε, γενικά τα τελευταία χρόνια τέτοιου είδους γνωμοδότηση ήταν το πράσινο φως, δηλαδή έλεγε το συνέδριο ότι το, το συνέδριο θεωρεί ότι εδώ έχουμε πιστή εικόνα των συναλλαγών της ε, Κομισιόν και της, ε, και της εικόνας της γενικής στο τέλος της χρηματοοικονομικής, συγγνώμη, της οικονομικής περίοδου της χρήσης και επίσης, και όπως επιτάσσει η συνθήκη, μια γνωμοδότηση όσον αφορά την κανονικότητα και το σύνομο των υποκειμένων συναλλαγών για αυτού του λογαριασμού. Όσον αφορά αυτό το δεύτερο είδο γνωμοδότηση, όσον αφορά την ομιμότητα και την κανονικότητα μέχρι σήμερα, αλλά και και ε, για το 2009 και για το 2010 το Ελληνικό Συνέδριο πρόκειται ε, να δώσει αρνητική γνωμοδότηση όσον αφορά την νομιμότητα και κανονικότητα αυτών των υποκειμένων συναλλαγών ανέκαθεν. Ε, καλά θα μπορούσαμε να προβληματιστούμε, αλλά προς το παρόν ε, με η εφαρμογή της συνθήκης πάντοτε οδηγεί σε δύο είδη γνωμοδοτήσεων. Μία επί των λογαριασμών, δηλαδή όσον αφορά τον ισολογισμό και ε, τους λογαριασμούς εκμετάλλευσης ε, και άλλη μία όσον αφορά νομιμότητα και κανονικότητα των υποκειμένων συναλλαγών. Και ανέκαθεν η δυσκολία ήταν όσον αφορά την γνωμοδότηση για την ε, νομιμότητα των υποκειμένων συναλλαγών και η κατάσταση αυτή συνεχίζεται. Προ λίγο συζητήθηκε το θέμα ε, των ταμείων συνοχής. Είναι ακριβώς ο τομέας όπου το ποσοστό των σφαλμάτων ε, είναι το πιο υψηλό. Όμως Επίσης έχουμε υψηλό ποσοστό, αρκετά υψηλό τέλο πάντων, πάνω κάτω και αλλού. Και κατά μέσο όρο διαπιστώνει το ελεγκτικό συνέδριο ότι το ποσοστό των σφαλμάτων κατά μέσο όρο για όλους τους τομείς είναι πάνω από το 2% του ποσού των δαπανών. Αυτό δε το 2% είναι το κατόφλι, το οποίο έχει καθορίσει το ίδιο ε, το συνέδριο για να αποφασίσει για το κατά πόσο θα δώσει ε, τη θετική γνωμοδότηση ή ου. Εάν επομένω το ποσοστό σφάλματο είναι κάτω από το 2%, τότε δίνει το πράσινο φω στο συνεδριό. Αν είναι πάνω, τότε δίνει αρνητική γνωμοδότηση. Το 2010 πάλι θα έχουμε ε, ελαφρώς ανώτερο του 2% ποσοστό ε, δηλαδή πάνω από το 2% και πάνω από το 2009. Αυτά. Okay, merci. The Commissioner, would you like to answer the... Κύριε Επίτροπε, θα θέλετε να απαντήσετε. Just to save some time. I, thought Α, για να μην χάνουμε το χρόνο μας, να σας πω, λέει ο κύριος Φιέλνερ. Πρώτα-πρώτα εισηγητής λέει και ο Πρόεδρος. Είχα ένα ερώτημα όσον αφορά το, το θέμα της συνοχής. Ήταν σαφής ερώτηση, αλλά δεν άκουσα να, μου απαντήσατε. Γιατί έχουμε αυτό το πρόβλημα όσον αφορά το Ταμείο συνοχή Να θέλετε να σας το ξαναδιατυπώσω. Γιατί είναι τόσο δύσκολο η DG Regio να τα καταφέρει. Καλά, μπορεί να είναι συνυπεύθυνα και τα κράτη-μέλη. Εντάξει. Όμως νομίζω ότι θα έπρεπε να μας πείτε κάπως περισσότερα. Πέραν το να μας λέτε για τη συνδιαχείριση. Τώρα, κάτι άλλο το οποίο ε, θεώρησε ότι ισχύει, αλλά το, το, το, το, το παρέλειψα. Μια τρόπο μιλάμε για τον εσωτερικό έλεγχο, την, ε, την έκθεση, για το 6 παράγραφος 3. Ωραία, όλα αυτά πρέπει να τα λάβουμε υπόψη και θα πρέπει να δούμε κατά πόσον είναι πραγματικά ιστορικό έλεγχο. Όμω, κάτι άλλο το οποίο είναι σημαντικό είναι το ότι τώρα έχουμε την περίληψη. 86 παράγραφος 4. 86 παράγραφος 4. Άρθρο 86 παράγραφος 4 και αυτό αφορά το ότι λαμβάνουμε τη μία έκθεση όταν λαμβάνουμε και την άλλη, τη συνθετική. Και ακριβώς τώρα έχουμε τα πρακτικά της συνεδρίασης που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την συνοπτική έκθεση. Οπότε μπορώ να διαπιστώσω ότι την Τετάρτη 1η 6 του 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει υπόψη αυτή την έκθεση 86 παράγραφος 4 σε σχέση με το 2010. Και εγώ αναρωτιέμαι γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν εμπόρεσε να εγκρίνει την περίληψη του 86-4 έγκαιρα πριν τη σημερινή συνεδρίαση. Γιατί αυτό θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Εντάξει, μπορούμε να συζητήσουμε για το σύνολο. Αλλά όμως θα μπορούσατε να έχετε εγκρίνει ε, αυτή την έκθεση. Κυρίως μια που ε, ανέκαθεν γινόταν έτσι. Και ξέρουμε το 86-3 εστάλει στο γενικό γραμματέα το Μάρτιο και πρώτη έκτου εσείς ε, ελάβατε υπόψη το κείμενο. Άρα είχατε αρκετό χρόνο ούτως ώστε σήμερα να έχουμε στα χέρια μας εγκεκριμένη σύνοψη και θα βοηθούσε πολύ. Ευχαριστώ. καλά, ευχαριστώ και δίνω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή στην κυρία Γκρέσλε. Σε μέτα. Σας ευχαριστώ. Πρώτα πρώτα. Για τις ε, του 64 είναι θέμα προϋπολογισμών. Ναι. Αργήσαμε σε σχέση με προηγούμενες χρήσεις. Ζητάμε συγγνώμη. Θα διορθωθούμε του χρόνου. Πάντως όπως και να έχει, έχει υποβληθεί η Ευρωπαϊκή έκθεση, οπότε και όταν έρθουμε εδώ για το, την ακρόαση του Δεκεμβρίου επί της απαλλαγής, θα είμαι έτοιμος τότε να συζητήσω ή αδίποτε ζητήματα που θεωρείται σημαντικά ότι πρέπει να συζητηθούν για το 86-4, για τις εκθέσεις μάλλον το 86-4. Τώρα, όσον αφορά τα της συνοχής, πρώτα πρώτα θα πρέπει να διαπιστώσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε σημαντικές δράσεις σε αυτόν τον τομέα στα πλαίσια τα, τα νομικά τα ισχύοντα. Οπότε, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις αρμοδιότητες που έχουμε, ε, περιοριζόμαστε, έχουμε όρια. Και αυτό είναι ένα από τα θέματα τα οποία μας προβληματίζουν σοβαρά. Και για αυτό ακριβώς στο, στο καινούργιο νομοθετικό πλαίσιο προτείνουμε να υπάρχει σημαντική αναβάθμιση των αρμοδιτών της Επιτροπής. Και αυτή η αναβάθμιση επίσης θα μας δώσει τη δυνατότητα να ασκήσουμε πίεση επί των πρώτων μέλων για να επιφέρουν τις αναγκαίες βελτιώσεις σε διαχείριση και έλεγχο. ώστε έτσι να αντιμετωπιστούν όλα τα σχετικά προβλήματα. Και έχουμε το θέμα των διαγωνισμών, των δημοσίων συμβάσεων, όπου ακριβώς πηγάζουν τα περισσότερα λάθη. Βλέπετε μας ότι έχει εδώ πέρα δύο όψεις αυτό το νόμισμα, ότι από τη μία πλευρά θα πρέπει να απλωστεύσουμε τις διαδικασίες και αυτό θα αποτελεί τμήμα των προτάσεων εις τη νέα οδηγία περί διαγωνισμών και προμηθειών και από την άλλη μεριά θέλουμε αυτές τις διατάξεις να τις θωρακίσουμε εναντί λαθών και να είναι και σαφής. Άρα εμείς περιμένουμε τώρα Θέλουμε αναμονή τέλο πάντων του νέου νομοθετικού πλαισίου. Άρα θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο την κατάσταση όσον αφορά την συνοχή. Και θα πρέπει να κινηθούμε στο ισχύον πλαίσιο. Και φαντάζομαι όλοι συμφωνείτε ότι δεν είναι τόσο εύκολο να επιφέρει κανείς αλλαγές πριν το τέλος της περίοδου προγραμματισμού να βρίσκονται δηλαδή κάποιες λύσεις που να μπορούν να ισχύσουν από τώρα και να είναι και αποτελεσματικές και, και οδηγούμεθα εις εντατικοποίηση κάποιων μέσων πολιτικής που να είναι συμβατά με τον νομικό πλαίσιο στον δηλαδή τη διακοπή και αναστολή των πληρωμών στον αγορά τους επιτόπου ελέγχους που είναι πάρα πολύ σημαντικά ως μέσα πολιτικής. Το πλαίσιο αυτό σχεδόν διακοπές των πληρωμών. Όλα αυτά θα πρέπει να συμφωνήσουμε πριν ανανεώσουμε τις πληρωμές για να δούμε τι δυνατότητες υπάρχουν επί τόπου ελέγχων, ελέγχου των εγγράφων. Αλλά όλα αυτά βέβαια μας φέρνουν επιπλέον, επιπρόσθετα έξοδα. Άρα θα είμαστε πολύ προσεκτικοί. Να, επομένω πώς είναι στην πραγματικότητα η κατάσταση. Και ο Επίτροπος Χαν θα έρθει στο Κοινοβούλιο για την ακρόαση που αφορά την πολιτική συνοχή, γιατί αυτός είναι ο άμεσα αρμόδιος. Και θα σα εξηγήσει ακριβώς τι κάνει για τα προβλήματα τη συνοχή. Thank you. σας ευχαριστούμε. Κυρία εισηγητρία. Κύριε εισηγητή, μάλλον στον κύριο Φιόνιο, Εσεί για να κλείσετε συζήτηση. Ναι, να ευχαριστήσω το συνέδριο, διότι ε, είπαν ότι στην ετησία έκθεση θα μα δώσουν αυτό που είπαν. Δηλαδή, θα μα ξεκαθαρίσουν πώ βλέπουν τι εκθέσει αυτέ. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ θετικό και θα πρέπει να διαβάσουμε τα έγγραφά τους για να ξεκαθαριστεί ο ορίζοντας, το τοπίο. Νομίζω τώρα είναι η κατάλληλη συγκυρία για να τα εξετάσουμε όλα αυτά. Να ανατρέψουμε σε αυτές τις δύο εκθέσεις και να δούμε κατά πόσον αποτυπώνουν με ακρίβεια την πραγματικότητα και να μην αφήνουν περιθώρια στο να αεροποιεί η Κομισιόν την κατάσταση. Άλλα δύο θέματα. Θα πρέπει να επανελθούμε στα θέματα της συνοχής. Και θα ήθελα να ε, ευχαριστούμε τον κύριο Σεμέτα για σε μας εξήγησε για το πώς θα ασκήσουν πίεση τα κρατη με τη διακόπη των πληρωμών γιατί φαίνεται σόφρον αυτό να μην δούμε, μόνο το θέμα της διακοπής, να δούμε και τα της ανάκτησης αυτής και, και πώς θα έχουμε και εκεί έλεγχους, διότι θα πρέπει να ξέρει η Κομισιόν ότι ο λόγος για την διακοπή έχει ε, εξεταστεί, έχει ληφθεί υπόψη και έχει διορθωθεί το πρόβλημα για να μην κάνουν συνέχεια τα την την να μην είναι υπότροπα. Οπότε όλα αυτά πρέπει να τα δούμε στη διαδικασία τη απαλλαγή, γιατί όπω προείπα, είναι πάρα πολύ σημαντικό το τι κάνει ο κάθε επίτροπο. Και άλλο. Είμαι σίγουρο ότι θα επανέλθουμε κατά την διαδικασία τη απαλλαγή τα είπε η κυρία Γκρέσλο, όσον αφορά τα μέσα τη χρηματοδότηση. λέγω ότι ακόμα δεν έχω καταλάβει όλα αυτά τα μέσα, τα αριθμιστικά, τα πούμε, financial engineering. Να δούμε όμως τι γίνεται όσον αφορά τις, ε, τις χρεοπιστώσεις, τους λογαριασμούς, τι έγινε αφού έκλεισε λογαριασμό στο Κοινοβούλιο και τώρα έχουμε νέους λογαριασμούς. Εγώ φαντάζομαι ότι όλα αυτά είναι νοικοκυρεμένα πλευρά λογιστικής και νομικής. Όμως και μόνο το ότι κάτι πρέπει να γίνει ε, είναι, σημαίνει ότι θα πρέπει να δούμε πιο λεπτομερώς κατά την διαδικασία της απαλλαγής και γι' αυτό παρακαλώ όλοι οι συναδελφοί να κάνουν αυτό που κάνω και εγώ να προσπαθήσουν να καταλάβουν τι τρέχει για να είναι αποδοτική η συζήτηση για όλα αυτά και να δούμε τι γνώμη θα διαμορφώσουμε για Τη ενέργεια τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής. Πάντως ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διότι κάλλιο αργά παρά ποτέ όσον αφορά την ε, περίληψη του εσωτερικού ελέγχου. Και σας υπόσχομαι όταν επανέλθετε τον Δεκέμβριο θα έχουμε και πάνω σε αυτό ερωτήσεις. Θα μπορούσα να προετοιμαστώ για τη σημερινή συνεδρίαση, αλλά τέλος πάντων ε, το ότι μας δίνεται την έκθεση λίγο πιο αργά δεν σημαίνει ότι θα ασχοληθούμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ εγώ, λέει ο πρόεδρο, και τώρα νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε αυτό το θέμα σήμερα στη διάταξη. Τώρα, το επόμενο βήμα στη διαδικασία θα γίνει τον Νοέμβριο. Οπότε και το ε, συνέδριο θα μα δώσει την τελική του έκθεση. Οπότε και τότε θα δούμε τι θα γίνει του χρόνου. Πάμε τώρα. Στο επόμενο σημείο του υπαριθμών τέτοια συμφωνημερινή διάταξη που είναι αυτή η έκθεση 5 του 2011, ειδική έκθεση όσον αφορά το ελεγκτικό συνέδριο, όσον αφορά αυτό το πρόγραμμα ε, SPS, ούτω ώστε να μπορέσουμε να έχουμε χρηστή διαχείριση. Η ειδική έκθεση το καθεστώ ενιαία ενίσχυση. ΚΕΕ. Υγιή δημοσιονομική διαχείριση. Πρώτα όμω το λόγο ο εισηγητή. Σα ευχαριστώ. Θα ξεκινήσω Ε, λέγοντάς σας ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά περίπλοκο θέμα καταρχήν, αλλά πρόκειται για 27 δις ε, ευρώ στην ουσία, δηλαδή για ένα σημαντικό κομμάτι του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Θα ξεκινήσω λέγοντας σας, ε, μάλλον ξεκινώ από το Ευρωπαϊκό, από το Ελληνικό Συνέδριο και να ευχαριστήσω τον κύριο Βερτάχη μόνο για την εκθεσή του, αλλά και για το πνεύμα συνεργασίας το οποίο κυριάρχησε. Το ίδιο να πω και προς την Κομισιόν, ο Επίτροπος Τσόλος, ε, δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτή την υπόθεση και να ευχαριστήσω και την γραμματεία της Επιτροπής μας. Πιστεύω πως αυτή η έκθεση της, ε, του ελεγκτικού συνεδρίου φτάνει την κατάλληλη στιγμή. Την επόμενη Τετάρτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει τις προτάσεις της για τη νέα γεωργική πολιτική και πιστεύω και κατάλαβα μάλιστα και από πλευρά του Επιτρόπου πως υπάρχουν κάποιες συστάσεις από πλευρά του ελεγκτικού συνεδρίου που θα λεφθούν υπόψη στις προτάσεις αυτές. Πιστεύω πως υπάρχουν δύο σημαντικά πράγματα, δύο σημαντικές επικρίσεις σε σχέση με το ναι, ναι, το, πρόγραμμα νέων πληρωμών ε, όσον αφορά τους ε, γεωργούς, ε, τους δικαιούχους, ε, τις, τι τις αγροτικές τα κτλ. Έχετε παραδείγματα γιές που δεν πρέπει να θεωρούνται γεωργικές αλλά που παρόλα αυτά αποτελούν αντικείμενο σημαντικών επιδοτήσεων. Το ίδιο και για τους ε, γεωργούς που δεν είναι πλέον ενεργοί αλλά που εξακολουθούν να παίρνουν σημαντικά ποσά από πλευράς των Βρυξελών. ίδια λογική ισχύει και για άλλα στοιχεία της ΚΑΠ τη κοινή πολιτικής πολιτική. Το ελεγκτικό συνέδριο είχε κάνει μια έκθεση όσον αφορά την γεωρική πολιτική και το περιβάλλον. Κάποιες φορές είναι τόσο αόριστες οι διατάξεις που τα χρήματα δεν φτάνουν εκεί που θα έπρεπε να φτάνουν. Μιλάμε για σχεδόν 29 δις ευρώ ετησίω. οπότε οι επικρίσεις αυτές δεν είναι αβάσιμες. Το πρώτο που μπορούμε να επικρίνουμε είναι ότι υπάρχουν πολλά δυνατότητες, πολλά πρότυπα στα διάφορα κράτη-μέλη, πολλά μοντέλα. Υπάρχουν πάνω από 20 και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η Κομισιόν ανέφερε μια ολόκληρη σειρά περιφερειακό, ιστορικό και στα κρατημέλη υπάρχει μια ευελιξία η οποία επιτρέπεται ώστε να είναι δυνατή η εφαρμογή αυτού του συστήματος. Η συνέπεια είναι πως τα κράτη-μέλη εφάρμοσαν το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης με το δικό του τρόπο το καθένα και οι ευρωπαϊκοί στόχοι που έχουν τεθεί ε, βρίσκονται σε κίνδυνο λόγω αυτής της κατάστασης. Κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα λάβει υπόψη βέβαια από αυτές τι επικρίσεις. Δεν χρειάζεται βέβαια να προκαταβάλουμε τη συζήτηση, θα το συζητήσουμε αργότερα, αλλά εγώ θα επιμείνω στις συστάσεις που διατυπώνω προς την κατεύθυνση της ε, Κομισιόν, ελπίζοντας ότι θα τις λάβει υπόψη. Καταρχήν, να σας πω ότι το καθεστώς ε, της ε, ενιαίας ενίσχυσης θα, είναι πολύ, θα πρέπει να είναι πολύ πιο καλά στοχοθετημένο. Αυτό σχετίζεται με την, το γεγονός ότι πρέπει να συνδεθούν μάλλον θα πρέπει να βρεθούν οι γεωργοί οι οποίοι δεν είναι πλέον στην παραγωγή και που δεν θα πρέπει πλέον να λαμβάνουν οποιαδήποτε ενίσχυση. Η απάντηση της Κομισιόν σε αυτό είναι ότι σύντομα θα έχουμε πρόβλημα με το πλαίσιο του ΠΟΕ. Ε, εντάξει, είναι πρόβλημα αυτό, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να αποφύγουμε να βρεθούμε σε κατάσταση... Ε, ανεπίλητη. Δεν μπορούμε να διατηρούμε δηλαδή αοριστίες στους ορισμούς μας, γιατί διαφορετικά κινδυνεύουμε να δίνουμε τα χρήματα στον κόσμο που δεν πρέπει να τα παίρνει. Αυτό είναι ένα, μια σύσταση την οποία θα πρέπει να τη λάβει σοβαρά υπόψη η Κομίσιον. Θα πρέπει να προσεγγίσει τα πράγματα διαφορετικά. Είτε στο πλαίσιο του ΠΟΕ να προσπαθήσει να βρει μια λύση ή, ε, ε, ή τότε, και εκεί το θέμα είναι ευρύτερο, να προσεγγίσει με ευρύτερο τρόπο τη χρήση των ε, γεωργικών ταμείων. Έπειτα, κατά τη διάρκεια τη περασμένη περίοδου φάνηκε ότι της επταετίας δηλαδή που μόλις περάσαμε, ε, ε, Υπήρξαν απρόβλεπτα προβλήματα. Υπήρξαν δηλαδή ε, λήψεις στην νομοθεσία και η Κομισιόν δυσκολεύεται να καλύψει αυτά τα νομοθετικά κενά. Και στο έγγραφο εργασία μου ε, προτείνω να δεθεί περισσότερη ε, εξουσία ε, στην Κομισιόν για να υπάρξει μια πραγματική νομική βάση για να συμπληρωθούν τα κενά. Αυτή τη στιγμή είναι εξαιρετικά περίπλοκη η κατάσταση. Όλα τα κρατημέλη πρέπει να ενεργήσουν προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί διαφορετικά τα χρήματα θα καταλήγουν σε λάθος χέρια. Για να μην γίνεται πλέον αυτό, θα πρέπει η διαδικασία να είναι πολύ πιο σαφή και ξεκάθαρη, έτσι ώστε η Κομισιόν να μπορεί να ελέγχει ακριβώ τι συμβαίνει. Κάτι ακόμα και εδώ ακολουθώ τη συμβουλή του ελεγκτικού συνεδρίου. Πρέπει να απλοποιηθεί περισσότερο το σύστημα και δεν χρειάζεται να επιμείνω περισσότερο σε αυτό. Κάτι ακόμα που θέλω να αναφέρω είναι ότι το ισχύον σύστημα εστιάζεται στους ήδη υπάρχοντες γεωργούς και είναι δύσκολο για τους νέους γεωργούς να εισέλθουν στην αγορά λόγω τον ιστορικό, του ιστορικού συστήματος, γιατί βασιζόμαστε σε αυτό που υπήρχε στο παρελθόν και από τη στιγμή που εμφανίζεται νέος Γεωργός δεν μπορεί εύκολα να έχει πρόσβαση σε όλα αυτά. Για τους νεοεισερχόμενους λοιπόν Γεωργούς υπάρχουν τεράστιες δυσκολίες και θα έπρεπε ένα σύστημα να χρησιμοποιηθεί που να είναι πολύ πιο δυναμικό και κατά συνέπεια θα πρέπει να υπάρχουν ε, επαρκή κίνητρα για την καινοτομία στον ιερικό τομέα, κάτι το οποίο δεν ισχύει σήμερα. Δύο σημαντικά θέματα λοιπόν. Οι νεοεισερχόμενοι δεν μπορούν εύκολα να έχουν πρόσβαση στην αγορά και επίσης δεν υπάρχουν αρκετά κίνητρα για την καινοτομία. Τέλος, να κάνω και μια γενικότερη φύσης παρατήρηση και να θίξω έτσι και ένα σημαντικό ζήτημα. Όταν βλέπουμε πώς λειτουργούν τα πράγματα, τα κάτι μέλη ζητούν όσο γίνεται μεγαλύτερη ευελιξία. Λένε ότι υπάρχουν μεγάλες αποκλήσεις στο κάτι μέλη, ακόμα και στο εσωτερικό των κρατών μελών και επιθυμούν η ευελιξία να ισχύει και για την εφαρμογή αυτών των ενιαίων ενισχύσεων, αλλά επί τη βάση της έκθεσης του συλλεκτικού συνεδρίου και ε, επί τη βάση της έκθεσης για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της γεωργίας και βλέπουμε και τον τρόπο με τον οποίο καταβάλλονται ε, ποσά σε λάθος ανθρώπους. Υπάρχει μια ασυναρτησία σε σχέση με αυτό που εμείς βάζουμε στόχο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό που τελικά εφαρμόζουν τα κράτη-μέλη. Εντάξει, ναι, μεν ευελιξία, αλλά πραγματικά έχω την αίσθηση πως ανεύθυνα χρησιμοποιούν αυτή την αρχή τη ευελιξίας στα κρατη Είναι σκληρά τα λόγια μου, ναι, αλλά επί τη βάση αυτών των τριών εκθέσεων του ελεκτικού συνεδρίου μπορούμε να πούμε πως τα κρατη παίζουν το παιχνίδι των Γιώργων και δεν ε, βλέπουν ποια είναι η πραγματική κατάσταση των ε, ίδιων αυτών ε, των Γιώργων για να δουν κατά πόσο αυτοί αντιστοιχούν στα κριτήρια που έχουμε ορίσει. Δηλαδή τα κράτη-μέλη φαίνεται να ενδιαφέρονται περισσότερο για την απόκτηση όσο γίνεται περισσότερων κονδυλίων από την Ένωση παρά για το τι θα γίνουν μετά αυτά τα χρήματα και αν θα πάνε στα σωστά χέρια ή όχι. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, είναι ένα ζήτημα το οποίο οπωσδήποτε θα πρέπει να το προσέξουμε. Σήμερα μιλάμε με το ελεγκτικό συνέδριο και με την Κομισιόν, θα, θα μιλήσουμε για τον τρόπο με τον οποίο ε, θα πρέπει να εφαρμόζεται το καθεστώς των ενιών ενισχύσεων για το πώς λειτουργεί και νομίζω πως ήταν και πολύ ενδιαφέρον να το συζητήσουμε αυτό και με τα κράτη-μέλη. Και εδώ δεν ε, έχω στο στόχαστρο το Συμβούλιο γιατί θα έχουμε την Προεδρία και θα έχουμε μια γενική συζήτηση που δεν θα εστιάσει στον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να εφαρμοστεί το σύστημα στα κρατημέλη και ότι θα έχουμε δυσκολίες όσον αφορά τη λειτουργία της Επιτροπής Ελευθερικού Ελέγχου. Πιστεύω ότι εκεί που έγκυται το μεγαλύτερο πρόβλημα στην εφαρμογή των κανόνων είναι τα ίδια τα κρατημέλη και είναι δύσκολο να ε, αγγίξουμε την ε, πληγή γιατί θα έχουμε αμέσως έναν υπουργό από ένα κράτος μέλος που θα μπορεί, ε, εύκολα να μας μιλήσει για τα μεγάλα προβλήματα εκτέλεσης όλων αυτών των προγραμμάτων αλλά θα ήθελα πραγματικά να γίνει μια τέτοια άμεση συζήτηση. Σας ευχαριστώ και Πρόεδρε, ευχαριστώ και το Ελεγκτικό Συνέδριο για την έκθεση αυτή και για την ε, γεωργική πολιτική γενικότερα. Είναι επικρίσεις σωστές και δίκαιες και να ευχαριστήσω και την Κομισιόν για τον αξιοσύνη σημείο, Το τρόπο με τον οποίο συνεργάστηκε μαζί μου. Είμαι πολύ περίεργος να δω πώς θα αντιδράσουν οι συνάδελφοι της Επιτροπής στις συστάσεις που διατύπωσα. Σας ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ. Θέλετε κάτι να πείτε από αυτού. Βεβαίως, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ που με καλείτε να σας παρουσιάσω την ειδική έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου μετά την παρουσίαση που έκανε ο εισηγητής σας και με την οποία συμφωνώ νομίζω ότι το καλύτερο για μένα θα ήταν να σας δώσω ορισμένες διευκρινήσεις σχετικά με ορισμένες παρατηρήσεις που έχει κάνει το ελεγκτικό συνέδριο με ορισμένα πιο τεχνικά στοιχεία δηλαδή με τις κριτικές τις οποίες εξίσχυσε ε, το συνέδριο εις ε, το ισχύον σύστημα των πληρωμών και το λέγω για να ε, επανακαθοριστούν οι στόχοι ε, της κοινή γεωργικής πολιτικής μετά το 2013 που είναι κάτι που προβλέπεται για την ενιαία πληρωμή όπως εκτελείται αυτή τη στιγμή. Για να είμαι σύντομος θα συγκεντρώσω τις παρατηρήσεις μου σε ε, τρία βασικά θέματα. Το πρώτο θέμα και το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι η νομοθεσία σχετικά με το καθεστώς της ενιαίας ενίσχυσης ε, η οποία ισχύει τώρα δεν συνάδει με τους στόχους κινήκτρων για γεωργική παραγωγή και για στήριξη του, του μεμονωμένου εισοδήματος των γεωργών. Και αυτό το αναφέρω σε δύο σημεία που υπάρχουν ασυνέπειες καταρχήν όσον αφορά την διατύπωση και δεύτερον την εφαρμογή στα κράτη-μέλη αλλά όσον αφορά την ευρωπαϊκή ε, ρύθμιση. Αυτή τη στιγμή η ευρωπαϊκή νομοθεσία προβλέπει ότι η ενιαία ενίσχυση περιορίζεται στα άτομα τα οποία έχουν δικαιώματα και ε, είναι, εξασκούν μία δραστηριότητα γεωργική σε επιλέξιμες περιοχές και ε, ο κάθε ένας από αυτούς τους όρους, επιλέξιμη γη, γεωργός, γεωργική δραστηριότητα, γη στη διάθεση του γεωργού, έχουν ερμηνευθεί κατά τρόπον ώστε ο κύκλος των δικαιούχων να έχει διευρυνθεί πέραν των ενεργών γεωργών που ήταν ο αρχικός στόχος της κοινή γεωργικής πολιτικής. Γι' αυτό και υπάρχουν ε, νέοι δικαιούχοι οι οποίοι δεν υπήρχαν ε, στο παρελθόν στις άμεσες ενισχύσεις. Οι νέοι αυτοί δικαιούχοι, των οποίων δεν υπάρχει γεωργική δραστηριότητα ή αποτελεί μόνο ένα μικρό μέρος της δραστηριότητος και ε, δέχονται ενισχύσεις διότι έχουν ε, κάποια ε, ακίνητη περιουσία. Και αυτό το έχει αναφέρει το ελεγκτικό συνέδριο στα προηγούμενα του, στις προηγούμενες εκθέσεις για τα αεροδρόμια, για τους σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, για τους δήμους που έχουν δημόσια πάρκα και υπάρχουν και νέοι καινούργοι ε, δικαιούχοι οι οποίοι είναι επενδυτές που δεν ενδιαφέρονται καθόλου για τη γεωργική εκμετάλλευση αλλά ψάχνουν ε, αποδοτικές ε, επενδύσεις ε, οι οποίες εξασφαλίζονται με αυτό το σύστημα. Η νομοθεσία λοιπόν δημιούργησε μία αγορά των δικαιωμάτων πληρωμής το οποίο ε, η οποία είναι διαφορετική από αυτό που υπήρχε στο παρελθόν. Και θα σας αναφέρω ένα πολύ γλαφυρό παράδειγμα το οποίο εξηγεί πολύ σωστά την κατάσταση. Ε, και αυτό το παράδειγμα το αποκομίζω από την έκθεση την οποία σας έχω υποβάλει. Ένας δικαιούχος το 2008 ε, απέκτησε για 200.000 ευρώ δικαιώματα πληρωμής ε, χωρίς όμως τη γη. Δηλαδή αγόρασε μόνο τα δικαιώματα και όχι τη γη που του εγγυώνται ένα εισόδημα πέραν του ενός εκατομμυρίου ευρώ για μία πεντιετία μέχρι να τελειώσει η τωρινή περίοδος της ΚΑΠ, δηλαδή μέχρι το 2013. Για να μπορέσει να δραστηριοποιήσει τα δικαιώματα αυτά, ο επενδυτής πρέπει να έχει και γη. Για να έχει λοιπόν ε, γη έχει ε, νοικιάσει ε, για 8.000 ευρώ το χρόνο μάλλον για 8.000 ευρώ για 45 βοσκοτόπους κακής ποιότητος που βρίσκονται σε κάποια ορεινή περιοχή πολύ μακριά από την μόνιμη κατοικία του. Για να διατηρήσει όμως σε καλή κατάσταση γεωργική αυτές τις εκτάσεις συμφώνησε με έναν κτηνοτρόφο ο οποίος βόσκει τα κοπάδια του σε αυτή την περιοχή. Οπότε μία επένδυση 200.000 ευρώ έχετε μία επένδυση ενός εκατομμυρίου που είναι μία πολύ καλή επένδυση εφόσον αποδίδει το πενταπλάσιο. Πολλοί επενδυτές θα ήθελαν να έχουν μία τέτοια απόδοση ε, και οι ίδιοι και σταματώ με αυτό το παράδειγμα. Το δεύτερο επίπεδο είναι στην εφαρμογή της νομοθεσίας από τα κράτη-μέλη. Οι εθνικές αρχές έχουν ε, μεγάλη διακριτική ευχέρεια για να εφαρμόσουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία και αυτές ε, οι εφαρμοστικές μέθοδοι πάντοτε δεν είναι προς της γεωργικής παραγωγικότητας που διαφέρει πολύ από το ένα κράτος στο άλλο και δεν βοηθά πάντοτε ε, την ε, γεωργική παραγωγικότητα. Παραδείγματο χάρη, σε ορισμένα κράτη υπάρχουν τελείως περιθωριακές ε, εκτάσεις που δεν είναι δυνατόν να καλλιεργηθούν ή δάση που θεωρούνται σαν κατά περίπτωση βοσκότοποι και καθορίζονται σε, ορισμένες, ορισμένα κράτη-μέλη ε, σαν επιλέξιμες εκτάσεις ενώ δεν ισχύει το, η ίδια συλλογιστική σε άλλα κράτη-μέλη. Είναι λοιπόν περίεργο πόσο έχει διευρυνθεί ο όρος επιλέξιμη έκταση ε, πέραν του λογικού. Δηλαδή υπάρχουν ε, δάση που δεν μπορούν να συγκριθούν με τις εκτάσεις όπου μπορεί κανείς να καλλιεργήσει σιτηρά. Και δεύτερον, για να μπορέσει κανείς να επωφεληθεί της ενισχύσεως θα πρέπει ε, η ε, εκτάσεις αυτές να είναι σε καλή περιβαλλοντολογική κατάσταση. Και αυτή, η, ε, αυτός ο ορισμός καθορίζεται από τα κράτη-μέλη και σε πολλές χώρες δεν σημαίνει τίποτα, για να μην σας πω απολύτως τίποτα. Υπάρχουν δηλαδή εκτάσεις οι οποίες βρίσκονται μέσα σε φυσικά πάρκα ε, και οι διοκτήτες ε, είναι δικαιούχοι νέων ενισχύσεων χωρίς να αναλαμβάνουν καμία δραστηριότητα ενώ στον ε, εσωτερικό, ε, στο προηγούμενο σύστημα δηλαδή στις άμεσες ενισχύσεις δεν επρόκειτο να λάβουν τίποτα. Βλέπετε λοιπόν ποια είναι η πρώτη διαπίστωση του ελεγκτικού συνεδρίου σχετικά με την αδικαιολόγητη αύξηση των δικαιούχων των ενιαίων ενισχύσεων. Δεύτερο θέμα, στην, ε, στο τωρινό σύστημα υπάρχει μία εσωτερική αντίφαση στις ενιαίες ενισχύσεις διότι αφενός θέλει να στηρίξει ε, το εισόδημα των γεωργών αλλά η ε, η ενίσχυση κατανέμεται χωρίς να ληφθεί υπόψη η μεμονωμένη κατάσταση κάθε ε, δικαιούχου ο οποίος ε, εκμεταλλεύεται τη γη του. Δηλαδή, καταρχήν συνδέεται με την επιφάνεια την οποία εκμεταλλεύεται, δηλαδή οι ενισχύσεις παραμένουν όπως το προηγούμενο σύστημα και κατανέμονται σε ένα μικρό αριθμό μεγάλων δικαιούχων. Θα αναφέρω τέσσερις αριθμούς πολύ ε, κραυγαλαίους, δηλαδή το 2009 0,4% των δικαιούχων έλαβαν 13% της συνολικής αξίας των πληρωμών, δηλαδή περίπου 100.000 ευρώ ανά δικαιούχο. Ενώ το 84% των δικαιούχων έλαβαν 27% 10% της συνολικής αξίας των πληρωμών, δηλαδή λιγότερο των 10.000 ευρώ ανά δικαιούχο. 100.000 από τη μια πλευρά και 10.000 από την άλλη. Υπάρχει λοιπόν ένα πρόβλημα κατανομής της μάζας του όγκου των ενισχύσεων. Μετά, η ενίσχυση η οποία χορηγείται ε, στο καθεστώς ενιαίων ενισχύσεων δεν αντικατοπτρίζει ούτε το κόστος της διατηρήσεως σε καλή κατάσταση των ε, ε, γεωργικών εκμεταλλεύσεων, το οποίο εάν, εάν συγκρίνουμε την κατάσταση στη Γαλλία ή σε μια περιοχή την οποία γνωρίζω πολύ και είναι εύκρατη και ε, σε μια ορεινή περιοχή το κόστος διατηρήσεως δεν είναι το ίδιο. Ούτε ε, το κόστος της αξίας ε, των υπηρεσιών που εκτελούνται από τους γεωργούς οι οποίοι διατηρούν διατηρούν το τοπίο και διατηρούν και πληθυσμό σε μια περιοχή η οποία θα ερήμωνε διαφορετικά. Τέλος, τρίτο σύστημα, το σύστημα των ενιαίων ενισχύσεων δίνει πολλές επιλογές στα κράτη-μέλη για την εφαρμογή του. Δηλαδή υπάρχουν περίπου 20 ε, συστήματα για να εφαρμοστεί η ενιαία ενίσχυση. Δεν θα σας απαριθμίσω και τα 20 αλλά ένα που είναι το ουσιαστικό και είναι το ιστορικό πρότυπο το οποίο εφαρμόστηκε από 11 ε, εκ των 17 κρατών μελών και στο πρότυπο αυτό το ποσό το οποίο ε, ε, καθορίζεται για τα δικαιώματα καθορίζεται από το ποσό που έπαιρνε στην περίοδο αναφοράς της τριετίας 2001 2003 στο παρελθόν δηλαδή αυτό το ποσό καθορίζει το δικαίωμά του για κατανομή ανα εκτάριο στην τωρινή περίοδο. Όσο όμως περνάει ο χρόνος τόσο αυτό το ποσό ε, διαφέρει από τις πραγματικές συνθήκες παραγωγής όπου οι νέοι γεωργοί οι οποίοι δεν είχαν δραστηριότητα ε, προδεκαετίες δηλαδή στην περίοδο αναφοράς εάν θέλουν τώρα να εγκατασταθούν σαν ε, γεωργοί πρέπει να αγοράσουν τα δικαιώματα πληρωμής αυτό αποτελεί ένα φραγμό για την ανανέωση του επαγγέλματος και την είσοδό τους. Δεν θα επανέλθω στις συστάσεις ε, του ελεγκτικού συνεδρίου διότι αυτές απορρέουν ακριβώς από αυτές τις παρατηρήσεις και ο εισηγητής σας τις ανέφερε αλλά δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω εδώ. Αλλά προφανώς αυτές οι συστάσεις γίνονται αυτή τη στιγμή από το ελεγκτικό συνέδριο για να ληφθούν υπόψη όταν θα ανακαταρτιστεί η κοινή γεωργική πολιτική για την περίοδο μετά το 2013. Δεν θέλω όμως να ε, ε, κλείσω χωρίς να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εργασία που έκανε ακολουθώντας το πνεύμα του ελεγκτικού συνεδρίου και το καλό κλίμα το οποίο είπε τις ε, σχέσεις μας και τις συζητήσεις μας μαζί του. Ευχαριστώ. Να ακούσουμε τώρα το σχόλιο της Επιτροπής. Ε, εντυπωσιαστήκαμε από αυτά που μας είπε και το ελεγκτικό συνέδριο. Παρακαλώ πρώτα η Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου καταρχήν να συγχαρώ εσάς για την ε, πρόσφατό σας διορισμό και να σας ε, ευχηθώ καλή επιτυχία στη νέα σας θέση. Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι Ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι, και εγώ θα ήθελα, θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τόσο το ελεγκτικό συνέδριο όσο και τον εισηγητή σας, τον κύριο Κερμπράντη, για τις παρατηρήσεις τους και τις συστάσεις τους. Όλα αυτά είναι πολύτιμες ε, συμβολές τον κοινό μας στόχο της περαιτέρω βελτίωση του, του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης όπως το έχουμε και να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις της σημερινής Ευρωπαϊκής Γεωργίας και φυσικά οι συστάσει του ελεκτικού συνεδρίου έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην προετοιμασία της μεταρρύθμισης που έχουμε ενώπιον μας και την οποία θα υιοθετήσει η Κομισιόν και θα δημοσιεύσει και τις προτάσεις της για την μεταρρύθμιση της ΚΑΠ μέχρι το 2020. 14 με 20. Χωρίς τώρα να αποκαλύψουμε όλες τις λεπτομέρειες της νομοθετικής πρότασης, θα ήθελα να τονίσω κάποια ζητήματα που ανέφερε τόσο ο κύριος Κερμπράντη όσο και ο κύριος Κρετά. Θα ήθελα να τονίσω ότι φυσικά η Κομισιόν γνωρίζει τα προβλήματα που έχουν υπάρξει και ελπίζουμε πως έχουμε κάνει ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών καταλήλως. Να ξεκινήσω με το πρώτο ζήτημα που είναι πολύ σημαντικό, αυτό που αποκάλεσε ο κύριος Γκερμπράντη, το θέμα των ορισμών. Εδώ έχουμε τον ορισμό του ενεργού γεωργού, την, την επιλέξιμη γη και την γεωργική δραστηριότητα. Και ο κύριος Κρετά μόλις ανέφερε κάποιες περιπτώσεις ακραίες, ας είμαστε ειλικρινείς, δεν είναι το φυσιολογικό που συμβαίνει όλη την ώρα ε, με βάση το συμμισχύον σύστημα, αλλά παρόλα αυτά θα πρέπει να αντιμετωπιστούν αυτές οι περιπτώσεις και να κλείσουν ή να διορθωθούν αυτές οι, αυτά τα παραθυράκια. Για τους τρεις σημαντικότερους ορισμούς που καθορίζουν την πρόσβαση στο σύστημα θα προτείνουμε νέους ορισμούς με πιο συγκεκριμένο τρόπο. Θα ήθελα όμως επίσης να πω, όπως το αναφέρατε και εσείς κύριε, κύριε Μπράντι, ότι επιμένουμε στην αρχή των αποσυνδεμένων πληρωμών. Θα ήταν πολύ πιο εύκολο αν λέγαμε ας πάμε πίσω στο παλιό σύστημα και να συνδέσουμε και πάλι τις πληρωμές μας με την παραγωγή. Αυτό φυσικά θα ήταν ο πιο στοχευμένος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να ανταποκριθούμε στα αυτά που είπε το ελεγκτικό συνέδριο για το πώς δηλαδή θα έχουμε ψηλότερη παραγωγικότητα. Αλλά μάθαμε από το παρελθόν ότι δεν είναι αυτός ο κατάλληλος τρόπος να προχωρήσουμε και γι' αυτό τουλάχιστον η Κομισιόν στην πρότασή της είναι αποφασισμένη να, να επιμείνει στις αποσυνδεμένες πληρωμές στην μεγάλη πλειοψηφία και έπειτα να προσπαθήσει να αντιμετωπίσει, και αυτό είναι πολύ περίπλοκο ζήτημα, να διατηρήσει δηλαδή την προσέγγιση της αποσύνδεσης αλλά και ταυτόχρονα καλύτερα να περιχαράξει και να ορίσει τις αρχές που δίνουν πρόσβαση στο σύστημα. Για τα διάφορα μοντέλα που αναφέρθηκαν εδώ να είμαι σαφής και εδώ η Κομισιόν θα, θα κάνει αυτό που ζητήσατε και εσείς και οι δύο έχουμε επίσης ε, καταλάβει ότι είναι και η ώρα να προχωρήσουμε προς ένα ενιαίο μοντέλο στην Ευρώπη που δεν θα βασίζεται στα ιστορικά στοιχεία πλέον, αλλά θα είναι πολύ κοντά σε αυτό που αποκαλούμε σήμερα το περιφερειακό μοντέλο. Το θέμα της ανακατανομής ανάμεσα στους γεωργούς. Ο κύριος Κρετέν σας έδωσε αυτό το μερίδιο των το πόσα παίρνουν διάφοροι δικαιούχοι. Και εδώ η Κομισιόν θα κάνει μια πρόταση για ένα πολύ πολύ σκληρό κανόνα οροφής. Κανείς δεν θα μπορεί να πάρει πάνω από ένα μάξιμο ποσό και θα υπάρχει μια σταδιακή μείωση των πληρωμών. Αυτό θα είναι ένα από τα κεντρικά μας στοιχεία για να μπορέσουμε να έχουμε πιο ε, αιτιολογημένα επίπεδα στήριξης εισοδημάτων και έπειτα. Καλύτερη στοχοθεσία των ε, πληρωμών. Αναφέρθηκε εδώ ότι δεν είναι σαφές για ποιο λόγο καταβάλλονται οι άμεσες πληρωμές. Ένα στοιχείο το οποίο θα εισαχθεί στη νέα μας πρόταση είναι το ε, πρασίνισμα, το greening της γεωργικής πολιτικής. Το 30% και αυτό ήδη αναφέρεται στα έγγραφα της Κομισιόν, το 30% των άμεσων πληρωμών θα πηγαίνουν άμεσα στα περιβαλλοντικά μέτρα. Και αυτό που είναι επίσης σημαντικό και για εσάς κύριε Κεμπράντη είναι ότι τα μέτρα αυτά είναι, ορίζονται σαφώς και ξεκάθαρα στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε εκεί η ευελιξία και το περιθώριο των κρατών μελών εδώ δεν, ε, είναι, δεν υπάρχουν σχεδόν, είναι σχεδόν μηδενικά σε σύγκριση με το μεγάλο ε, περιθεώριο ελιγμού που υπήρχε μέχρι τώρα. Καλύτερη στοχοθεσία επίσης γίνεται μέσω της πληρωμής που εισάγουμε για τους νέους, τους νέους εισερχόμενους γεωργούς που το ανέφερε και αυτό και ο Σκρατέν και αυτό επιπλέον των κανονικών άμεσων πληρωμών και της στήριξη που μπορούν να έχουν οι νέοι γεωργοί από το δεύτερο πυλώνα για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Αυτά είναι δύο παραδείγματα για το πώς μπορούμε να αποσαφηνίσουμε ότι επίσης βλέπουμε την ανάγκη για καλύτερη στοχοθέτηση των χρημάτων από ό,τι συμβαίνει τώρα. Κάτι ακόμα που είναι σημαντικό και για τον κύριο Γκερμπράντη και έχει δίκιο είναι ότι χρειάζεται να δοθούν περισσότερα χρήματα στην έρευνα και την καινοτομία. Και πάλι, αν δούμε το έγγραφο της ε, Κομισιόν για το, για το δημοσιονομικό πλαίσιο θα δείτε ότι τα χρήματα που έχουμε βάλει για το γεωργική καινοτομία και έρευνα έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Τώρα εμείς πρέπει να βρούμε το σωστό τρόπο ώστε να χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα αυτά για τα κατάλληλα προγράμματα. Αλλά συμφωνώ με το Συλλεκτικό Συνέδριο και με τον κύριο Μπράντι ότι υπάρχει χώρος να γίνουν πολύ περισσότερα σε επίπεδο εκμετάλλευσης όσον αφορά την έρευνα και την καινοτομία από ό,τι γίνεται μέχρι τώρα. Και έπειτα. Τώρα, κάτι ακόμα το οποίο ρώτησε και ανέφερε και ο εισηγητή είναι η ευελιξία των κρατών μελών. Και εδώ πρέπει να αναφέρουμε τα εξή. Ναι, κάποια ευελιξία είναι απαραίτητη για τα κράτη-μέλη, διότι δεν υπάρχει κανόνας ε, UNISEX για όλα τα κράτη-μέλη. Υπάρχουν ένα σωρό διαφορετικές δομές. Διαφορετικές δομές εκμεταλλεύσεων και συνθήκων εκμετάλλευσης. Είναι απαραίτητο λοιπόν να υπάρχει κάποιος χώρος ελιγμού για τα κράτη-μέλη. Αυτό όμως που μπορούμε να κάνουμε καλύτερα και εκεί όπου μπορούμε να κάνουμε περισσότερα είναι το πώς θα περιχαρακώσουμε, θα περιορίσουμε, θα ορίσουμε καλύτερα τα περιθώρια που αφήνουμε στα κράτη-μέλη. Και ως προς αυτό Καλωσορίζω όλος ιδιαιτέρως τη σύσταση του εισηγητή, του κύριου Γερμπράντη, που λέει ότι πολύ συχνά βλέπουμε μόνο την, στην εφαρμογή των κανόνων μας εκεί που υπάρχουν ε, τα κενά ή τα ελαττώματα. και οι νομοθετικές μας προτάσεις να γίνουν με τέτοιο τρόπο όπου υπάρχει δυνατότητα για εκχώρηση αρμοδιοτήτων στην Κομισιόν, ώστε η Κομισιόν να μπορέσει να δράσει πιο γρήγορα. Γιατί όπως έλεγα, οι κανόνες είναι περίπλοκοι. Τα κράτη-μέλη, όπως είπε και το ελεγκτικό συνέδριο, κάποιες φορές ε, δίνουν τη δική τους ερμηνεία για την εφαρμογή των μέτρων και εδώ η Κομισιόν χρειάζεται καλύτερη και πιο αποτελεσματικά εργαλεία από ό,τι αρχική διαδικασία που παίρνει δύο-τρία χρόνια μέχρι ότου μετά να διορθωθεί το πρόβλημα. Την Τετάρτη φέτο λοιπόν η Κομισιόν θα παρουσιάσει τι νομοθετικέ προτάσει και αν τι διαβάσετε προσεκτικά θα δείτε ότι πολλά, πολλά πραγματικά από τα όσα σύστησε το ελεγκτικό συνέδριο αλλά και ο εισηγητή με τι συστάσει του θα αντιμετωπιστούν. Και έπειτα θα πρέπει να συζητήσουμε αν είναι αρκετά όλα αυτά που θα προτείνουμε ή αν στη συζήτηση ανάμεσα μας αν θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο τα πράγματα ή όχι. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα να δώσω το λόγο στους ε, βουλευτές και κυρία, πρώτος, πρώτη κυρία Γκρέσλε. Να ευχαριστήσω το συνέδριο. Πολύ ωραία η έκθεσή σας. Ε, κύριε Κρετά, ε, σας ευχαριστώ και εκτιμούμε την ε, έκθεσή σας, αν και εγώ ίδια ακόμα προσπαθώ να καταλάβω ακριβώς τι τα κάνουμε όλα αυτά τα στοιχεία. Συνεχίζω γερμανικά. Ε, ευχαριστώ, αλλά εδώ αντιλαμβάνουμε ότι μιλάμε για το 1 τρίτο των των πληρωμών 30 δισεκατομμύρια ευρώ και γιατί έργησε τόσο η έκθεση αυτή γιατί νομίζω ότι έχει, αργήσει, έχει καθυστερήσει τέσσερα χρόνια έπρεπε να έχουμε ενημερωθεί πιο νωρίς για να επέμβουμε διότι αυτή τη στιγμή έκθεση έχει το πρόβλημα ότι δεν μπορούμε να επέμβουμε. Μπορούμε δηλαδή να προσβλέπουμε στις καλύτερες εποχές που ανέφερε ο Γενικός Διευθυντής διότι δεν πρέπει πάντοτε όταν έχουμε κακές εμπειρίες να ελπίζουμε ότι θα φτιάξουν τα πράγματα διότι η κατάσταση αυτή ήταν γνωστή το ξέραμε, το έχουμε συζητήσει επανειλημμένως και ε, ιδίω ε, λόγω της, ε, των κακών νέων από τον τύπο και γιατί αργήσατε τόσο πρωί πολύ, γιατί θα πρέπει να αλλάξουν οι κανόνες. Επίσης, ποια είναι η δικιά σας αξιολόγηση, διότι ουσιαστικά οι ενισχύσεις αυτές ε, αποβλέπουν στο να υπάρχει μία ανταγωνιστική γεωργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά έτσι η ε, γεωργία της Ευρώπης δεν είναι ανταγωνιστική και ε, ξέρω περί τίνος ομιλώ διότι τον Ιούλιο πήγαμε στην Ουγγαρία και είδαμε ότι το μέσο μέγεθος της εγκαταστάσεως γεωργικής είναι 2,5 εκτάρια και είπε η Επιτροπή ότι έτσι πρέπει να μείνει. Πού είναι λοιπόν οι μηχανισμοί για την κατεύθυνση ε, ε, ε, προς μια ανταγωνιστική γεωργία έπρεπε να, ε, γεωργίες, έπρεπε έχουμε και διάφορα προγράμματα ε, για την ανανέωση του επαγγέρματος γιατί η απερίμωση της υπαίθρου είναι σημαντική και έπρεπε να δώσουμε καλύτερες δυνατότητες στους νέους. Κάτι θα ήθελα να μου σχολιάσετε και από αυτού. Επίσης, η αποδέσμευση δεν σημαίνει άμεσα ότι ε, μπορούμε μόνο να ανατρέξουμε στο ιστορικό πρότυπο. Θα ήθελα να ξέρω τι άλλες ιδέες υπάρχουν. Δηλαδή αν πιστεύετε ότι αν στηρίξουμε τη δραστήρια γεωργία αυτό μπορεί να γίνει με το 30% ε, στη, στον τομέα αυτό ή θα πρέπει ο κανονισμός να ξαναλάξει; Ευχαριστώ. Δεν βλέπω κανέναν άλλον από τα κράτη-μέλη που θέλει να λάβει το λόγο και νομίζω ότι ο τελικός ομιλητής που πρέπει να επανέλθει είναι ο εισηγητής. Ξέχασα τον κύριο Ντί, με συγχωρείτε και του λέω να με συγχωρήσει. Ευχαριστώ τον εκπρόσωπο του ελεγκτικού συνεδρίου διότι ε, δεν ε, αναφέρομαι εδώ στο σύνολο αλλά αναφέρομαι σε συμπεριφορές τις οποίες ίσως δεν είχαμε προβλέψει αλλά βλάπτουν την Ευρωπαϊκή Ένωση διότι ο στόχος της αναθεώρησης το 2003 ήταν ακριβώς να αναθεωρηθεί η γεωργία της Ευρώπης και να συνάδει με ε, τον ΠΟΕ. Και όταν αφού μπαίνουμε στην τελική ευθεία των διαπραγματεύσεων επί τη βάση των προτάσεων της Κομισιόν, θεωρώ ότι αυτή η έκθεση παρά το ότι έφτασε αργά, έφτασε τελικά τη σωστή στιγμή. Και θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορούσαμε να το συντεριάσουμε με τον τζίρο, αλλά όμως μιλούμε για εισοδήματα γεωργικά. Όταν έχουμε μια κρίση που χτυπάει τα εισοδήματα, όπως είδαμε τα τελευταία χρόνια σε κάποιους ε, κλάδους, όχι παντού, σε κάποιους όπως ε, τα σιτηρά, αλλά τα είδα, το είδαμε στην κτηνοτροφία, αυτό θα πρέπει να συνδυαστεί όχι με το τζίρο, αλλά με το εισόδημα. Πολύ σωστό, γιατί βάλατε από τον τύπο τον είδα το δάχτυλο. The court the... Θα ήθελε το Ελληνικό Συνέδριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τα σχολιάσει αυτό το οποίο ελέγχθησαν. Από ό,τι φαίνεται όχι. Επομένως, τι λέει ο Ναι, λέει η Γραμματεία, ε, η... θέλουν, θέλουν να απαντήσουν. Άρα, δεν σα είδα. Ε, ο κύριος από το Συνέδριο, ναι πρόεδρε, μια πολύ σύντομη παρατήρηση το γιατί έφτασε αργά αυτό δυστυχώς. Είναι κλασικό το ότι όλες μας οι εκθέσεις φτάνουν εκ των υστέρων και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γι' αυτό. Για τον απλό λόγο ότι χρειάζεται κάτι επί το οποίο να γίνει έλεγχος οικονομικός και μετά να γίνει έκθεση. Το 2003 διαμορφώθηκε η νέα πολιτική, αλλά δεν υλοποιήθηκε παρά μόνο το 2005. Και αυτό το οποίο εγώ σας παρουσίασα είναι το αποτέλεσμα σειρά οικονομικών ελέγχων μεταξύ 2006 και 2010 σε 17 κρατημέλια. Επομένω, χρειάζεται κάποιος χρόνος. Αλλά, κάπως για να σχετικοποιήσουμε τα πράγματα, πρέπει να σας πω ότι κάποιες από αυτές τις πληροφορίες είχαν δημοσιευθεί σε κάποιες ε, επιμέρους εκθέσεις ή στο παρελθόν. Όμως η διαφορά είναι ότι αυτή τη φορά μπορέσαμε όλα αυτά να τα βάλουμε σε προοπτική, να εξαγάγουμε κάποια συμπεράσματα από αυτές τις ε, επιμέρους παρατηρήσεις επί των συναλλαγών που είχαμε ε, εξετάσει. Όμως δυστυχώς αναγκαστικά όλα αυτά βγήκαν αργά. Όχι υπερβολικά αργά ευτυχώς, ούτως ώστε να ληφθούν υπόψη από την Κομισιόν οι παρατηρήσει μα οπότε με την ευκαιρία σα ευχαριστούμε ε, για, για όσα είπατε κύριε εκπρόσωπο τη Κομισιόν. Πρόεδρο. Σα διαβεβαιούμε ότι αυτά που την υπόψη. Κύριε Ισηγητά, θέλετε το λόγο. Ναι, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόκειται για πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση να μπορούσε εκ των προτέρων να κάνει τον έλεγχο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ε, εκ των προτέρων υποβάλει τι εκθέσει επί τη βάση των όσων είπαμε. Θα δούμε μάλλον την Τετάρτη να μην επαναλάβω τα ίδια. Όμω τώρα ε, ε θα είναι μεγάλο επηρεασμό να χρησιμοποιήσουμε τα τη ΚΑΠ, αλλά τέλο πάντων δεν είναι εδώ χώρο ε, για τέτοια πράγματα γιατί αυτό το οποίο θέλουμε εδώ να κάνουμε είναι να βρίσκουμε τις αιτίε των πραγμάτων και κατά τη δική μου άποψη η γεωργική πολιτική είναι πολιτική συναισθηματικά φορτισμένη. Καταλαβαίνουμε τους λόγους όμως έτσι τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα. Είναι πολιτικές κάποιες επιλογές όπως αυτά που λέμε για την Ουγγαρία τα δραματικά για την καταστροφή. Τέλο πάντων, ε, ό,τι αποφασίζει, αποφασίζει το ελληνικό συνέδριο και άκουσα διάφορε και άλλε τέτοιε ριζοσπαστικέ προτάσει. Ε, πιο, πιο ριζοσπαστικέ. Να κάτσουμε με την κυρία Γκρέσσα να τα συζητήσουμε γιατί θα με ενδιαφέρε ε, η, ομάδα τη κυρία Γκρέσσα να με υποστηρίξει. Όμω, τέλο πάντων, έχω μία ερώτηση όσον αφορά τα προβλήματα που έχουμε εντοπίσει με τον ΠΟΕΑ. Νομίζω ότι βρισκόμαστε στο εξή αδιέξοδο, στο εξή φαυλοκύκλο. Θέλουμε πιο πολλά χρήματα, θέλουμε να αξιοποιούνται. Δεν μπορούμε να συνδέσουμε αυτά τα κονδύλια με την παραγωγή και αν τα συνδέσουμε με, με, την τα ιστορικά ποσά της ε, ε παραγωγής, τότε απομακρυνόμαστε πολύ και όλα αυτά μπορούμε να τα κατεβάσουμε στον ΠΟΕ. Όμω έτσι μετακινούμεθα προς ε, άλλο σύστημα. Αυτό είναι αυτονόητο και κατά τη γνώμη μου νομίζω θα πρέπει να εξασφαλίσουμε το ότι οι επιδοτήσει αυτές θα πηγαίνουν εκεί που χρειάζονται και όχι εκεί που θέλουν τα κράτη-μέλη. Εμένα κάπως με ανησυχεί το ότι εάν γίνουν αυτές οι αλλαγές πορείας σε κάποια χρόνια θα χρειάζεται νέα έκθεση, όπου πάλι θα πρέπει να δούμε πώς διατέθηκαν τα χρήματα, γιατί πήγανε σε μέρη που δεν έπρεπε να πάνε, οπότε τότε, εν κατακλείδη, ίσως θα έπρεπε να σας αναφέρω ότι όντως ε, νομίζω ότι θα μπορούσε να καταλήξει εκεί το ελληνικό συνέδριο να κάνει εξάντεκ των προτέρων προτάσει και εκθέσει. Θα, ναι, θα ακούσουμε τι θα υποθεί την Τετάρτη, λέει ο Πρόεδρο, γιατί θα είναι πάρα πολύ σωστό να έχουμε και κάποια γνωμοδότηση από την Επιτροπή Γεωργία. Ε, να μα πει τη γνώμη τη ε, Επιτροπή Γεωργία επί... επί των λέει Επιτροπή. Οπότε και εμεί αυτόν να ρωτήσουμε εμεί ω Επιτροπή την Επιτροπή Γεωργία. Καλοδεχούμενε στις συμβουλέ σα, κυρία Επιτροπή. Τώρα λοιπόν θα με τελειώσω στο σημείο 4 και πάμε στο σημείο 5. Το 5, το οποίο πάλι είναι μια ε, ειδική έκθεση του Ενεργητικού Συνεδρίου όσον αφορά ε, το, αν ήταν αποτελεσματικά τα συγχρηματοδοτηθέντα από το ΕΤΠΑ έργα στον τομέα του τουρισμού. Κύριε Βόν, ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα-πρώτα Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να μακρηγορήσω. Ε, έχετε δει, ελπίζω, και διαβάσει, συνάδελφοι, το δικό μου έγγραφο. Έχουμε τι αρχικέ πατρίδε και είδατε εδώ πέρα ότι πρόκειται για τον τουρισμό που είναι πάρα πολύ σημαντικό κλάδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε περίπου 100 εκατομμύρια θέσει εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα μπορούσατε ε, να διαπιστώσετε ότι έχουμε 4,6 εκατομμύρια ευρώ που προέρχονται από το ΕΤΠΑ από το, κατά την περίοδο 2006 και γι' αυτό και σας λέω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί του θέματος. Επίσης, συναδελφοί, θα είδατε στην έκθεσή μου τα σχετικά με εμβέλεια και στόχους του ελέγχου, τι είπε το συνέδριο, τι διαπίστωσε, γιατί αυτό το οποίο διαπίστωσε ήταν αρκετά θετικό, ε, είπε για... Ε, ε, το 73% συνόλου τη αύξηση τη με 4% δυναμικότητα υποδοχή, 58% θέση εργασία των έργων. Οπότε τώρα όμω προβληματίζεται το ελληνικό συνέδριο και προβληματίζεται και γιατί σε πολλέ περιπτώσει που μελετήθηκαν διαπιστώθηκε ότι η χρηματοδότηση δεν είχε εξαρτηθεί από τη δημιουργία θέσεων εργασία. Δηλαδή οι στόχοι δεν είχαν τεθεί στην αρχή του προγράμματο. Επίση ε, η εποπτεία και η αξιολόγηση δεν έγιναν ακόμα και όταν υπήρχαν κάποιοι στόχοι ευθύ εξ αρχή του προγράμματο και επίση το 2% των επιλέξιμων θεώρησαν ότι η συμμετοχή του ΕΤΠΑ έφερνε περισσότερη γραφειοκρατία ει βάρο του. Από πλευρά της απάντησης Κομισιόν θα μπορείτε να διαπιστώσετε στην έκθεση ότι η Επιτροπή απάντησε ε, περίπου στο ότι έχουμε συνδιαχείριση για αυτή την ε, πολιτική, την πολιτική συνοχής για στόχους, για την απλούστευση, ότι όλα αυτά είναι στόχοι και έχουν ε, ε, τεθεί σαφώ και πρόκειται να ισχύσουν και στο μέλλον. Όσον αφορά τώρα τι δικέ μου προτάσει ε, που περιέχονται στο τέλο περίπου τη εκθέσεω, λέω ότι είναι πάρα πολύ θετικά από όλα αυτά τα προγράμματα γιατί όντω δημιούργησαν θέσει απασχόληση και επίση συμφωνώ με το ότι είναι σημαντική αυτή η στόχη. Δημιουργούνται θέσει εργασία, ίσω είναι ο πιο σημαντικό στόχους. Επίσης λέω εδώ ότι έχουμε και άλλους στόχους που μπορούν να οδηγήσουν ε, στην ε, αύξηση της απασχόλησης μέσω του τουρισμού και ως παράδειγμα αναφέρω την αύξηση των επισκεπτών. Επίσης αύξηση των δαπανών των τουριστών και την ποιότητα, την αυξημένη ποιότητα υπηρεσιών και στέγασης. Όλα αυτά μπορούν να τονίσουν ε, την απασχόληση μέσω του τουρισμού. Επίσης συμφωνώ ε, και προτείνω ότι θα πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση ε, της διαδικασίας ε, επιχορήγησης του ΕΤΠΑ και η στοχοθέτηση να είναι καλύτερη από ό,τι στο παρελθόν. Θα γίνει περισσότερη προσπάθεια επίσης λέω ώστε να βρω την απλούστευση της επιχορήγησης. Πάντα το λέγαμε αυτό. Ανέκαθεν λέγαμε ότι η απλούστευση είναι πολύ σημαντική για τους επιλέξιμους του ΕΤΠΑ μπορούμε να σημειώσουμε πρόοδο και ίσως την επόμενο γύρο της ανθεώρησης των ταμείων να το κάνουμε αυτό. Ευχαριστώ το μικρό συνέδριο, αλλά ευχαριστώ και τη γραμματεία που βοήθησε. Αυτά, Πρόεδρε. Thank you. Then I would like to... Ευχαριστώ κύριε Βόν, ο Πρόεδρος. Ο κύριος Ισπριτό από το Ελληνικό Συνέδριο έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να έρθω εδώ, να παραστώ σε αυτήν την ανταλλαγή απόψεων επί τη βάση αυτού του εγγράφου που ε, περιέχουν την ειδική έκθεσή μας με υπαρθμόν 6 για το 2011 όσον αφορά την συγχρηματοδότηση. Να μην επαναλάβω προς τον κύριο Βον κάτι γιατί σημαντικά αυτό το οποίο είπε, αλλά έχει ολοκληρωθεί το έργο του. Αυτή η ειδική έκθεση υπαρχημών 6 ε, είναι η πρώτη μας έκθεση, η οποία 100% αφορά τον τουρισμό και την Αφορά κάποιες επενδύσεις. 2006 είναι η περίοδος που καλύπτεται. Μιλούμε για 4,6 δις ευρώ. Αυτά είναι χρήματα του ΕΤΠΑ. Κάναμε μια δειγματοληψία 26 προγραμμάτων από όλα τα κρατημέλη και θέλουμε να δούμε κατά πόσον αυτά βοηθούν τους στόχους. Τα κρατημέλη είναι βασικά όσον αφορά τα προγράμματα του τουρισμού. Αυτό αφορά τη διαχείριση. Υπάρχει εδώ το θέμα της επιγορικότητας και οι εθνικές αρχές μπόρεσαν έτσι να διαχειριστούν και να παρακολουθήσουν τα προγράμματα. Έγινε επιτόπου επίσκεψη και έλεγχος των ελεγκτών και έχουμε τα αποτελέσματα της έρευνας, σύμφωνα με τα οποία πολλά προγράμματα, μαρίνες, δρόμοι, τρένα, κάμπινγκ, μουσεία, μνημεία χρηματοδοτούνται υπό τον τίτλο «Τουρισμός». Γιατί υπάρχουν και εκπαιδευτικά κέντρα και άλλα τα οποία επίσης πρέπει να λυθούν υπόψη. Όπως είπε ο κύριος Βόν στον εργασίας, εμείς καταλήγουμε στο ότι υπήρχαν θετικά αποτελέσματα από όλα αυτά τα προγράμματα. Έχουμε αυτές τις συστάσεις, σύμφωνα με τις οποίες θα πρέπει τα προγράμματα να έχουν στόχευση στους στόχους και να διαπιστώνεται κάθε φορά κατά πόσο βοηθήσουν την ανάπτυξη αυτά τα προγράμματα και την απασχόληση. Εμεί συστήσαμε ότι θα πρέπει τελικά αυτά να θεωρούν καλέ πρακτικέ να τα ενθαρρύνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζουμε ότι είναι, έχουν καλή σχέση κόστος αποτελέσματο και θα πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει στόχευση για και με προτεραιότητα τον τουρισμό. Βλέπω με μεγάλη μου χαρά ότι ε, εδώ ε, στα συμπεράσματά του συμφωνεί μαζί μας ο κ. Βόν και τον ευχαριστούμε. Επίσης, μεγάλη μου χαρά βλέπω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε αυτό το ψήφισμα που λέει Ευρώπη νούμερο ένα τουριστικός προορισμός. Αυτά τα συζητήσαμε σε σχέση με τον έλεγχο. σε σχέση με τα πλαίσματα του ελέγχου και σε σχέση με τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου εδώ, σας αναφέρω το πόσο εγκάρσιο χαρακτήρα είναι ο τουρισμός, οριζόντιο χαρακτήρα τέλο πάντων. Ε, έχει παντού επιπτώσεις και όλοι οι κλάδοι πάλι έχουν επιπτώσει τον τουρισμό. Και γι' αυτό ε, έχουμε ιδιάζοντα χαρακτήρα των θέσεων ασχολούνται με τουρισμό, ότι είναι κάπως ευάλωτες. Όλα αυτά πρέπει να υπόψη από τοπικές αρχές και περιφερειακές αρχές. Όμως, η αναφορά μας και το ψήφισμα είναι στο τιμή σχήματος. Επομένως, θα πρέπει και η Επιτροπή να παίξει για την Επιτροπή Συνοχής σημαντικό ρόλο. Και πότε θα πρέπει να δούμε το ότι ένταλο ε, πρέπει να τεθεί και ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτή την πολιτική. Ευχαριστούμε, ο ο και η Κομισιόν έχετε το λόγο. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε και τον κύριο Βόν για την έκθεσή του, αλλά ευχαριστούμε και τον ίδιο συνέδριο διότι ε, διενήργησε αυτόν τον οικονομικό έλεγχο που εμείς χαιρετίζουμε και επίσης ε, συμφωνούμε με τα συμπεράσματα ε, από αυτόν τον έλεγχο που διαπιστώθηκε ότι η χρηματοδότηση του ΕΤΠΑ είναι πάρα πολύ σημαντική για τον ε, τουρισμό και επίσης θεωρούμε ότι είναι θετικά τα συμπεράσματα του ΕΤΠΑ. Έτσι θα έχουμε σαφέστερες θα φέρει στόχοθέτηση. Θεωρούμε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο ισχύει για όλη την πολιτική της συνοχής και είναι αυτό το οποίο και εμείς προτείνουμε γίνει στο μέλλον. Μια που διαπιστώθηκε ότι έχουμε τέτοιες ε, ανάγκες. Σύμφωνα με τα όσα είπαμε την περασμένη εβδομάδα. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό θα πρέπει να είναι η καρδιά προτάσεων για το μέλλον. Και θεωρούμε ότι αυτό θα πρέπει να χαρακτηρίζει όλη τη διαδικασία, ακόμα και στο τελείωμα του προγράμματος. Μα είπε για τις διαχειριστικές αρχέ ο κύριος Βον, για την επιλογή ε, των ε, επιδοτουμένων από το ΕΤΠΑ προγραμμάτων. Όμως θα πρέπει να έχουμε συγκεκριμένα κριτήρια όσον αφορά το τι θα επιλεγεί και τι θα τύχει στήριξη. Οπότε συμφωνούμε πάρα πολύ με αυτό το σημείο και θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει μεγαλύτερη συνάρθρωση των στόχων μεταξύ τους. Και έτσι είναι πιο αποτελεσματικό το πρόγραμμα. Και αξιολόγηση είναι καλύτερη. Έτσι γίνεται αξιολόγηση, αλλά έτσι θα γίνει πιο εύκολη. Όσον αφορά τώρα την υποστήριξη για τον τουρισμό, ξέρετε ότι το ΕΤΠΑ δεν δίνει ε, στον τουρισμό ε, κάθε αυτό, αλλά υποστηρίζουμε τις, περι... τις ε, στατικές περιοχές ανάπτυξης που κάποιες φορές καλύπτουν τον τουρισμό και το είδος της βοήθειας μπαίνει σε διάφορα προγράμματα ανάλογα με το αν μια περιφέρεια προσπαθεί κάτι να, πάθει, να πετύχει. Σίγουρα επενδύουμε σε αξιολόγηση. Ενθαρρύνουμε τα κρατημένα να κάνουν αξιολόγηση και να εστιάζονται στις αποτελεσματικές παρεμβάσεις. Οπότε και θα θέλαμε να δούμε πώς η χρηματοδότηση του ΕΤΠΑ στη διάφορες περιφέρειες έχει διάδραση με το τι γίνεται σε άλλες περιοχές και να δούμε. Επίσης θα πρέπει να επικεντρώσουμε ενδιαφέρον μας το πώς θα προσθέσουμε περαιτέρω την πρόσβαση στην ε, υποστήριξη του ΕΤΠΑ. και θέλουμε να γίνει απλούστευση του ισχυρού καθεστώτος για τους δικαιούχους. Και υπάρχει η απλούστευση βέβαια για τις διεύγειες αρχές, αλλά τελικά το πιο σημαντικό είναι οι δικαιούχοι και όχι αυτοί που διαχειρίζονται τα ταμεία και τους πόρους να είναι το επίγεντο της απλούστευσης. Σας ευχαριστούμε και πάλι. Ευχαριστούμε και τον κύριο Γον για τις ε, συστάσεις Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γκρέσλε έχει ζητήσει το λόγο. Η έκθεση είναι πολύ ενδιαφέρουσα ε, και θεωρούμε όλοι το θέμα του τουρισμού πολύ σημαντικό ε, και εάν δούμε τώρα τις ε, στατιστικές βλέπουμε ότι ε, υπάρχει ένα ποσοστό συμμετοχής. Ε, βλέπω ότι δεν υπάρχει τόσο πολύ ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία διότι αν κανείς έχει ε, ανοικοδομήσει και οροποιήσει ε, ε, το κτίριό του και κάνει ένα ξενοδοχείο πέντε αστέρων το οποίο βελτίωσε με πόρους Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρέπει να εξετάσουμε πού πηγαίνουν οι πόροι της Ευρωπαϊκής Ενώσεως διότι ε, το να έρχεται μία ομάδα ατόμων με ένα μακρύ ευχολόγιο και ε, να μπορούν να ε, ε, υποβάλουν προτάσεις δεν σημαίνει ότι θα πρέπει κανείς να τις δέχεται μετά από τα πορίσματα του ελεγκτικού συνεδρίου. Μπορούμε λοιπόν να δούμε πού βρισκόμαστε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω το συνέδριο για αυτές τις διαπιστώσεις και όλες αυτές οι εκθέσεις δεν ξέρω αν δίνονται σε όλους τους βουλευτές, αλλά είναι πολύ χρήσιμες ε, στο πλαίσιο των πολιτικών συζητήσεων που αρχίζουν για τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές. Μήπως ε, θα ήταν ε, η κατάλληλη στιγμή να γίνει μια ευρωπαϊκοποίηση αυτών των ευρωπαϊκών δημόσιων κονδυλίων να έχουμε μια ευρωπαϊκή πολιτική τουρισμού σύμφωνα και με το ψήφισμα που έχει μάλιστα ψηφίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε την τύχη να είμαστε ο πρώτος τουριστικός ε, προορισμός. Ε, μήπως λοιπόν θα πρέπει να τα παγιώσουμε όλα αυτά και μάλιστα εντυπωσιάστηκα από τον αριθμό ότι το 1 τέταρτο των φορέων θεωρούν ότι με η άνευ ενίσχυση θα είχαν ούτως ή άλλως υλοποιήσει το, το σχέδιό τους. Θα έλεγα ότι είναι η άρνηση εντάξει, όχι ίσω η άρνηση, αλλά θα πρέπει αυτό να μας κάνει να διερωτηθούμε για την αποτελεσματικότητα των δημοσίων δαπωνών. Ε, σύμφωνοι για την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, επίση σύμφωνοι για την απλοποίηση, χρήση χαρακτήρια στην εισηγητή μα. και να συγχαρώ και την Ουαλία για την ε, πολύ ωραία πρόσβαση στον ημιτελικό του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράγκμπι. Λοιπόν, άπαξ και ξεκίνησε η πτήση. Βλέπω ότι Τώρα τα προγράμματα του τουρισμού είναι ένα από τους τομείς που λειτουργούν πλέον αποτελεσματικά. Όταν βλέπω τα διάφορα προγράμματα εύχομαι και τα άλλα να μπορούσαν να λειτουργούν εξίσου καλά όσο ο τουρισμός. Παρόλο που και εκεί θα υπάρξουν προβλήματα στη χρηματοδότηση. Και έχω μία ερώτηση διότι ε, ε, δεν απάντησαν όλοι οι γιατί δεν απάντησαν όλοι οι υπεύθυνοι για τα προγράμματα. Ε, διότι εφόσον χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή ε, Ένωση θα μπορούσαν τουλάχιστον να απαντούν όταν τους κάνουμε κάποια ερώτηση. Γιατί δεν απάντησαν, υπήρχε κάποιο συγκεκριμένος λόγος για τον οποίο δεν απάντησαν και αν ε, δεν επαρκούν ε, οι λόγοι, τι έγινε, έγιναν εξαιρέσεις από το ελεγκτικό συνέδριο και επίσης όσον αφορά τις συστάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου για το αποτέλεσμα συμπράξεως ε, ή ότι χρειάζεται το πρόγραμμα οπωσδήποτε κάποια ενίσχυση είναι κάτι το οποίο μπορεί κανείς ε, εκ προημίου να επαληθεύσει ή ε, θα χρηματοδοτηθούν λιγότερα προγράμματα εάν και άλλα πρέπει να ε, χρηματοδοτηθούν. Θα ήθελα δηλαδή να ακούσω ποια είναι η θετική αξιολόγηση του ελεγκτικού ο συνεδρίου διότι αντιλαμβάνουμε τις επικρίσεις αλλά εξεπλάγει ότι λειτουργεί το σύστημα τόσο καλά και ε, ελπίζω ότι ο σημείο αυτό η Ευρω... Ε, τα κράτη της Ευρώπης αναλαμβάνουν ε, το κόστος της προσθεθμένης αξίας. Ευχαριστώ και θέλω να κάνω μία ερώτηση. στο λέγεται ότι χρησιμοποιήσαν 4 ε, ε, δισεκατομμύρια, πέραν των 4 δισεκατομμυρίων για το πρόγραμμα αυτό, το οποίο είναι πολύ σημαντικό ποσό και ότι η απορρόφηση ήταν 75% για την ε, δημιουργία θέσεων και στη σελίδα 19 λέγεται ότι δημιουργήθηκαν 220.000 άμεσες θέσεις εργασίας. Έγινε λοιπόν εστιασμός στο, στο τομέα ή εγώ παρανόησα τον αριθμό των θέσεων που δημιουργήθηκαν με όλα αυτά τα χρήματα. Θέλει κάποιος να προσθέσει κάτι στο τέλος. Τότε το δικαστήριο για να σχολιάσει. I'd like to thank uh, for your question. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ερώτησή σας και για το ενδιαφέρον σας για αυτή την έκθεση. Θέλω να τονίσω την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία για αυτά τα προγράμματα και να σας δώσω τις συστάσεις μας, τα εμπορίσματά μας ε, για και πώς αυτά θα ληφθούν υπόψη. Η σύστασή μας, ας πούμε, τονίζει την ιδέα ότι η αξιολόγηση της Επιτροπής για την επόμενη περίοδο to uh, undertake a evaluation of aid in this sector to consider the extent of which its former cost effective. Λέει ότι τα χρήματα αυτά θα πρέπει καλύτερα να στοχευθούν και τα λοιπά. Ο κατάλογος των σχεδίων θα μπορούσε να είναι πολύ κρίσιμος και σημαντικός. Αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι προσεγγίζουμε την ειδική μας έκθεση ελέγχοντας προγράμματα τα οποία έχουν ολοκληρωθεί στα κράτη-μέλη στη δειγματοληψία που κάναμε. Σε σχέση με τους διαχειριστές των προγραμμάτων, θα ήθελα να πω ότι είχαμε πάνω από 200 προγράμματα στην δειγματοληψία και αυτά αξιολογήθηκαν από το συνέδριο μέσω των απαντήσεων που έδωσαν στα ερωτηματολόγια. Θεωρώ λοιπόν ότι το δείγμα μας ήταν επαρκές για να φτάσουμε στα συμπεράσματα στα οποία καταλήξαμε. Μόνο τέσσερις δικαιούχοι δεν απάντησαν στα ερωτηματολόγια μας. I'd like to add the idea of the uh, combine our recommendation. Θα ήθελα να προσθέσω ότι θα πρέπει να συνδυαστούν τα πορίσματα αυτά τη έκθεση με το ψήφισμα του Κοινοβουλίου, διότι το ψήφισμα αυτό δίνει μια ευρύτερη εικόνα για το τι σημαίνει ο τουρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση. I think, uh, uh, document, our document, our working, uh, the uh, uh, working document could consider, could be considered good. Νομίζω πως αυτό το έγγραφο εργασίας θα πρέπει να εξεταστεί από την Κομισιόν ώστε να σκεφτεί και να σχεδιάσει την επόμενη περίοδο σε σχέση με αυτά τα θέματα. About, uh, employment. Because, uh... Σε σχέση με την απασχόληση, γιατί κατάλαβα ότι πολλά χρήματα δαπανήθηκαν για αυτές τις δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του 2006 μέχρι 10 και μόνο 2.560 θέσεις απασχόλησης δημιουργήθηκαν. Όμως πιστεύω πως αυτοί οι δείκτες δεν είναι οι κατάλληλοι, διότι η ιδέα δεν ήταν να δημιουργηθούν θέσεις πάνω απ' όλα, Η ιδέα ήταν να καταλάβουμε και να γίνουν καλά προγράμματα για αυτή την περίοδο και με, σε ποιο βαθμό μπορούσαν να βελτιωθούν αυτά τα προγράμματα και αυτές οι πολύ σημαντικές δραστηριότητες. In our discussion in the court during the audit and during uh, uh, το συμπέρασμά μας λοιπόν είναι ότι δεν είναι πολύ θετικά τα αποτελέσματα όσον αφορά την απασχόληση και τη δημιουργία νέων θέσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε αντίθεση με τα τεράστια ποσά που δαπανήθηκαν γι' αυτά. Αλλά στην παράγραφο 32. Κοιτάξτε, δεν έχουμε πολύ χρόνο, διακόπτει ο Πρόεδρος. Σε περίπτωση που έχετε πολύ συγκεκριμένες απαντήσεις για τις ερωτήσεις που ετέθησαν και τις παρατηρήσεις που έκαναν ε, οι βουλευτές σας, θα ήθελα αυτές να τις, διαπα... κάνετε με σύντομο τρόπο, γιατί στις 6 έχουμε μια άλλη συνεδρίαση και ήδη έχουμε ξεπεράσει το χρόνο μας. Θα ήθελα να δώσω το λόγο και στην Επιτροπή ΔΕ Εάν έχετε λοιπόν κάποιες συγκεκριμένες και σύντομες απαντήσεις να δώσετε, δώστε τις, αλλά όχι επί μακρόν. Παρακαλώ. I think it's necessary to, to give some uh, additional information if it's necessary for this. Αν χρειάζεται θεώρηση, μπορώ να σας πω μερικές παραπάνω πληροφορίες από αυτού, αλλά... Um, presentation, uh, uh, point of view of my team. Αλλά εδώ πέρα βλέπω τι μου λένε για αυτόν τον ε, έλεγχο οι συνεργάτε μου. Ο μιλητή μιλά μακριά από το μικρόφωνο και ακούγονται τα μισά από λέει. I εάν έχετε συγκεκριμένε απαντήσει, παρακαλώ ε, μπορείτε να τι διαβάσετε απευθεία στα στα μέλη του Κοινοβουλίου που, που, που ενέχονται σε αυτό. Ε, μάλιστα, έχετε το λόγο, Κομισιόν. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να σα πω είναι ότι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρήσαμε ότι τα αποτελέσματα αυτού του οικονομικού ελέγχου ε, ε, ε έδωσαν κάποια θετικά αποτελέσματα για επενδύσει, για τουρισμό και σε σχέση με τα αποτελέσματα αυτών των επενδύσεων σε αυτά τα προγράμματα, διότι κάποια από αυτά τα αποτελέσματα ήταν ακόμη καλύτερα από όσα παίρνουμε από άλλες, από άλλες επενδύσεις ε, αυτό το Ιωνία Απόβαρο επίση ήταν καλύτερο από τους άλλους κλάδους. Ε, επίσης, στην περιφερειακή πολιτική νομίζω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη κατα... κατάτμιση των ε, πόρων και αυτό το έχουν διαπιστώσει μια σειρά τη αξιολογία. Επομένω, αυτό το οποίο για το μέλλον είναι να εστιάσουμε στα αποτελέσματα και επίση να υπάρχει μεγαλύτερη συγκέντρωση των πόρων Γιατί θα πρέπει να υπάρχει μια κρίσιμη μάζα με βασική διάρθρωση όσον αφορά τους στόχους της πολιτικής που θέλουμε να πετύχουμε και ε, η χρηματοδότηση να πηγαίνει απευθείας εκεί που, θεωρούμε ότι επιτυγχάνονται οι στόχοι. Επομένως να βρεθεί ένας μηχανισμός που να αποσπάσει περισσότερο από για το μέλλον τώρα σε σχέση με το ότι θέλουμε να έχουμε περισσότερα στοιχεία για την αποτελεσματικότητα ε, του, του, της στήριξης του τουρισμού έχουμε μια μεθοδολογία αξιολόγηση που επενδύουμε τώρα και λέμε ότι θέλουμε αξιολόγηση των επιπτώσεων του τύπου counterfactual, δηλαδή να μην συνδέεται με τα πραγματικά περιστατικά. Επομένως αυτό να δούμε. Ότι αυτό θα πρέπει κάπως να γίνει ε, όχι, να γίνει σε, σε συγκεκριμένο πλαίσιο και όχι πανευρωπαϊκά. Γι' αυτό και διστάσαμε να αναδεχθούμε αυτό που είπε το Ελληνικό Συνέδριο, να τα κάνουμε όλα εμεί. Γιατί νομίζω θα πρέπει να είναι υπευθυνότητα με περιφέρειε, κρατημέλη κλπ. Και εκείνοι επομένω να ανακάθονται και να αξιολογούν το πώ αυτοί αξιοποίησαν του πόρου. Το τελευταίο που θα σα αναφέρω είναι το ότι οι θέσει απασχόληση που άμεσα δημιουργήθηκαν, μην ε, ξεχνάτε ότι αυτή η στατιστική ήταν ε, επί τη βάση δείγματο και όχι από τη βάση όλων των προγραμμάτων. Άρα πάμε για ψηλότερη απόδοση. Και έχουμε επίση και αποτέλεσμα έμεση δημιουργία θέσεων απασχόληση, γιατί ε, επομένω μπορεί κανεί να έχει ω στόχο όχι μόνο θέσει απασχόληση να έχει, το να αυξηθούν οι επισκέπτε, οπότε και αυτό ε, βοηθάει έμεσα οι επιχειρήσει που δεν συνδέονται άμεσα με τα χορηγούμενα κεφάλαια, του χορηγούμενου πόρου. Αυτά. Ε, Εμεί ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρο, και τώρα θα ολοκληρώσει ο εισηγητής Βον. Θα είμαι λακωνικός, αν όχι τηλεγραφικός. Κύριε Χολμαϊό, ρώτησε γιατί με μερικοί δεν απάντησαν στο ερωτηματολόγιο. Ξέρω εγώ μπορεί να είναι διακοπές. Τόσο πολύ μπορεί να βόηθαγε ο τουρισμός. Ήταν διακοπές και δεν απάντησαν στο ερωτηματολόγιο. Κύριε Χολμαϊό, επίσης, ο κύριος Σοντή, είπε το θέμα της κάτι για την προσθετικότητα, πάρα πολύ καλά μας τα είπε ότι όντως πέραν της έρευνας θα προχωρούσε το πρόγραμμα και χωρίς την κοινοτική χρηματοδότηση. Για την προσθετικότητα επίση να μην ξεχνούμε ότι και οι στόχοι της πολιτικής και η στόχοι 2020 είναι ανάπτυξη και απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και από την έρευνα αυτή προκύπτει ότι η χρηματοδότηση στον τουρισμό βοηθάει σε όλα αυτά. Ακριβώς και γι' αυτό είπαμε ότι θα πρέπει να εκταμιεύονται χρήματα από τα ταμεία για τον τουρισμό. Φυσικά και είμαι υπέρ αυτών των συστάσεων του συνεδρίου. Ευχαριστώ συνάδελφοι για το όσα είπατε. Ελπίζω να αξιοποιήσουμε αυτή τη συζήτηση όταν συζητήσουμε στο μέλλον και για την απαλλαγή, αλλά και όταν συζητάμε και για τα ταμεία. Πρόεδρο, σα ευχαριστούμε. Νομίζω ότι ολοκληρώσαμε με αυτό το σημείο σήμερα τη διατάξεω. Θα συνεχίσουμε επομένω αύριο το πρωί στι 9. Ακριβώ. Σα ευχαριστώ.